Good morning. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους λέει στα γαλλικά ο πρόεδρος. Δίας. Και στα ισπανικά καλημερίζει. If you want to take your seats. Αν θέλετε καθίστε παρακαλώ. Thank you for your silence. Ευχαριστώ που είσαστε ήσυχοι και ήρεμοι. Καθίσατε. Ξεκινάμε με το δεύτερο εργαστήριο αυτού του σεμιναρίου που διαρκεί δύο ημέρες σε αυτή τη συνάντηση την διακοινοβουλευτική της Επιτροπής μας για την δημοκρατική λογοδοσία στον χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και, ε, ε, ασφάλειας. Ξεκινάμε με το επόμενο πάνελ. Έχουμε εδώ τους εκπροσώπους του για αυτή τη συνεδρίασή μας που θα διαρκέσει μία ώρα και 15 λεπτά και έχουμε την παρουσία ανάμεσά μας με ιδιαίτερη τιμή του κυρίου Άλετ Βίλιαμς, πρόεδρο του Συλλογικού Σώματος της Eurojust. Τον καλωσορίζουμε θερμά. Την κυρία Ρενάτε Βέβερ, συνάδελφό μας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ, στην, Ευρωπαϊκή, στην Ευρωβουλή, που είναι η συγγήτρια σε σχέση με το Eurojust όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο αυτό, και την κυρία Κριστίν Ντεφρένιε, που είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βελγικής Γερουσίας. Ξεκινάμε λοιπόν. Και δίνω τον λόγο αμέσως στον κύριο Αλέντο Βίλιαμς, πρόεδρο της Eurojust. Παρακαλώ. Um, very much, Σας ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι Εθνικών Κοινοβουλίων, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση να σας προσφωνήσω σήμερα το πρωί. Προτίθεμαι να ακολουθήσω τους όρους της πρόσκλησης και σύντομα να αναφερθώ σε δύο πτυχές. Πρώτα, τις ε, ενεξελίξει οι δραστηριότητες τη Eurojust και δεύτερον για το μέλλον τη Eurojust, ιδιαίτερα για το θέμα της αξιολόγησης και τη δημοκρατικής λογοδοσία τη Eurojust. Στρέφομαι στο παρόν πρώτα. Η Eurojust λοιπόν, η αποστολή της επιβεβαιώθηκε στη συνθήκη της Λισαβόνας και αυτή η αποστολή είναι να υποστηρίζει και να ενδυναμώνει τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ερευνητικών και διοκτικών αρχών σε περιπτώσεις σοβαρών διασυνοριακών εγκλημάτων. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι στο οποίο εργαζόμαστε από τότε που δημιουργήθηκε η Eurojust το 2002. Και αν δείτε τους αριθμούς των περιπτώσεων που εξετάσαμε, σωστό είναι να πει κανείς νομίζω ότι είμαστε σχετικά επιτυχείς, αρκετά επιτυχείς Είχαμε 200 αναφορές από τα κράτη-μέλη στο παρελθόν. Το 2009 είχαμε περίπου 1.400 τέτοιες ε, περιπτώσεις ε, που ζητήθηκε συνδρομή από τα κράτη-μέλη από την Eurojust. Είναι επταπλάσια η αύξηση αυτή που σημειώθηκε στον όγκο εργασίας μας και το κάνουμε αυτό φυσικά με περιορισμένα κονδύλια και πόρους. Είμαστε μια, ένας μικρός οργανισμός, έχουμε ένα προϋπολογισμό 30 εκατομμυρίων ευρώ έχουμε στο διοικητικό επίπεδο περίπου 200 στελέχη, 200 άτομα. Υπηρετούν 50 διοκτικές αρχές και από τα 27 κράτη-μέλη. Και έχουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο διοργανώνουμε περίπου 130 συναντήσεις για την εξέταση τέτοιων περιπτώσεων κατά την διάρκεια ενός έτους. Στόχος τέτοιων συναντήσεων είναι να αντιμετωπιστούν δυσκολίες στην αντιμετώπιση στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, ιδιαίτερα δυσχερών περιπτώσεων. Αυτό που κάνουμε είναι μια απλή, προσφέρουμε ένα απλό και μη γραφειοκρατικό εργαλείο για τις εθνικές διοκτικές αρχές. Ένας εισαγγελέας, ένα κράτος μέλος, μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να στείλει ένα email και να έρθει σε επαφή έτσι και έχοντας επαφή με, με, με την εθνική εκπροσώπηση των εθνικών διοκτικών αρχών, η Eurojust <coughs> μπορεί να δει και να διαπιστωθεί ότι 4-5 άλλα κράτη-μέλη εμπλέκονται. Μπορεί να περάσει κανεί στο διάδρομο να μιλήσει με του 4-5 αρμόδιους και να έχει μια συνάντηση συντονισμού όπω την αποκαλούμε για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Τα προβλήματα υπό το εθνικό πρίσμα μπορούν να θεωρούνται αξεπέραστα. Πώς μπορούν να συντονιστούν έρευνες, πώς μπορούν να μοιραστούν πληροφορίες με 5-6 κράτη-μέλη. Πώ μπορεί κανεί να διασφαλίσει ότι θα παγώσουν τραπεζικοί λογαριασμοί στη σωστή χρονική στιγμή. Πώ μπορεί να διασφαλίσει κανεί την εκτέλεση των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψη. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία επιλύουμε εμεί στην Eurojust και τα αντιμετωπίζουμε και προσφέρουμε τι υπηρεσίε μα ώστε οι κοινέ ερευνητικέ ομάδε να μπορούν να λειτουργούν. Δίνουμε και τα κονδύλια που διασφαλίζουμε για την λειτουργία αυτών των κοινών ε, ομάδων. Και αυτό είναι ένα κίνητρο για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματο. Στι δικέ μα περιπτώσει, όπω θα ανέμενε κανεί, αυτέ αντλούνται από τις περιπτώσεις που δυσχεραίνουν και τη ζωή και δημιουργούν προβλήματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Λαθρεμπόριο ναρκωτικών, λαθρεμπόριο ανθρώπων, κάθε είδους ε, τρομοκρατίας, ε, πράξη τρομοκρατίας ε, και κυβερνοεγκλήματος με διασυνοριακές πτυχές που συνδέονται στις δραστηριότητες αυτές. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τους εταίρους μας στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα με τη Europol. Έχουμε την έδρα μας στη Χάγη, όπως και η Europol. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση εργασίας με τη Europol, την Europol και όπως ανέφερα και πιο πριν, ανέφερα τις 130 περιπτώσεις συναντήσεων από πλευράς μας. Η Europol παρακολουθεί ένα τρίτο περίπου αυτών των συναντήσεων στην Eurojust. Σας παρουσίασα έτσι με αδρές γραμμές μια σκιαγράφηση εν συντομία των ε, δραστηριοτήτων μας. Θέλω να στραφώ στο μέλλον της Eurojust τώρα. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και είναι μια θέμα και είναι μια ιδιαίτερα με μεγάλες προκλήσεις συνδεδεμένη περίοδο στο μέλλον αυτό. Τώρα έχουμε τη νέα απόφαση, η αναθεωρημένη απόφαση για τη Eurojust όπου απαιτούνται τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2011 σε αυτή την απόφαση αναδιάρθρωσης. Και η κατεύθυνση αυτής της απόφασης είναι η Eurojust να είναι το δυνατόν όσο περισσότερο λειτουργική και αποτελεσματική. Υπάρχουν διάφορες πτυχές πτυχέ σε αυτά. Δεδομένου του ότι ο χρόνος πιέζει θα αναφέρω μία πτυχή και είναι ίσως η πιο κέρια και κύρια για την ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι σαφώ αυτό ένα ιδιαίτερα θέμα η Eurojust. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε να συνδράμουμε τα κράτη-μέλη και τα σώματα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκή Ένωση στην καταπολέμηση σοβαρών <clears throat> διασυνοριακών εγκλημάτων πρέπει να παίρνουμε την πληροφορία, τις πληροφορίες σε έγκαιρο χρόνο ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Και σύμφωνα με το άρθρο 13 τη νέα απόφαση, υποχρέωση καθορίζεται για τα κράτη-μέλη να παράσχουν αυτές τις πληροφορίες στην Eurojust. Κυρίως για οποιαδήποτε περίπτωση σοβαρού εγκλήματος με διασυνοριακή διάσταση που θα εμπλέκει και την, το αίτημα συνδρομής και αρρωγής σε σχέση με τα κράτη-μέλη προς την Eurojust. Και έχουμε επίση και μια πρόταση η οποία θα αρχίσει να ισχύει τον Ιούνιο 2011 του χρόνου για ένα εθνικό σύστημα συντονισμού. Αυτό σημαίνει ότι πραγματικά θα υπάρχει μια, ένα γραφείο της Eurojust που θα λειτουργεί σε κάθε κράτος μέλος θα συναποτελείται, θα συναπατίζεται από επαείοντες στην δικαστική συνεργασία. Θα εξετάζουν να βλέπουν αν είναι οι περιπτώσει αυτέ ενδεδειγμένε για τι αρμοδιότητε τη Eurojust ή μήπω αν θα πρέπει στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο να αναφέρονται. Υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα και εγχειρήματα τα οποία αναπτύσσονται και βρίσκονται σε εξέλιξη σαν αποτέλεσμα τη συνθήκη Λισαβόνα. Δεν έχω χρόνο παρά μόνο να αναφέρω κάποια από αυτά σε αυτή τη φάση. Ίσως θα έπρεπε να αναφέρω την συμμετοχή της Eurojust στην Επιτροπή για την Εσωτερική Ασφάλεια COSI, στο COSI. Συγγνώμη, ναι, σας ευχαριστώ. Ε, πήγαινα πολύ γρήγορα, έτσι, ναι, επειδή πιέζει ο χρόνος, γι' αυτό έτρεχα. Ωραία, θα επιβραδύνω λίγο. Γνωρίζοντας ότι πιέζει ο χρόνος, όπως έλεγα. Λοιπόν, όπως έλεγα, για το COSI, εμείς στην Eurojust ελπίζουμε ότι μπορούμε να παράσχουμε, αν θέλετε, δικαστικές προτάσεις και κίνητρα όσον αφορά την, κυρίως την προοπτική επιβολής του νόμου και σεβασμού του νόμου σε σχέση με την κόζη. Κάνοντας αυτό και προβλέπουμε ότι θα γίνεται αυτό με τους συνδέσμους μας με το άτυπο διαβουλευτικό συμβουλευτικό φόρουμ, το βήμα των Γενικών Εισαγγελέων που ξεκίνησε ή προσεγγίστηκε υπό την Ισπανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα ακολουθείται ως πρωτοβουλία από τη Βελγική Προεδρία και την χάνει συνέχεια. Θα διοργανώσουμε την επόμενη συνάντηση αυτού του φόρουμ που σε αυτό συνέρχονται οι ε, γενικοί εισαγγελείς, ε, διευθυντές γενικών εισαγγελιών από τα κράτη-μέλη το Δεκέμβριο του 2010. Ε, Φέτο θα γίνει αυτή η σύνοδος. Μια άλλη σαφώς σημαντική πτυχή για μας είναι οι, προ... οι προτάσεις για κανονισμούς υπό το άρθρο 85 τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε ότι ελπίζει ότι θα υποβάλει μια πρόταση για αυτού τους κανονισμούς το 2012. Και αυτά νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή κλίματος και περιβάλλοντος για την Eurojust και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό θεωρώ όπως απαιτεί η συνθήκη να υπάρχουν προτάσεις, ιδέες, input σε σχέση με τις αρχές της αναλογικότητας, της επικουρικότητας και τα λοιπά που πρέπει να είναι σεβαστές όταν θα αρχίσουν να λειτουργούν βέβαια και να σχεδιαστούν, θα σχεδιαστούν και θα τεθούν υπό έγκριση αυτοί οι κανόνε και κανονισμοί. Ήδη στη Eurojust εξετάζουμε τι διαφορετικέ εναλλακτικέ δυνατότητε που είναι διαθέσιμε. Κάναμε κάτι το οποίο πιστεύω ήταν ένα ενδιαφέρον σεμινάριο στην Bruges του Βελγίου 20-22 Σεπτεμβρίου, κάποιες λίγες εβδομάδε πιο πριν δηλαδή και ενδιαφέροντα σεμινάρια έγιναν. Ένα τέτοιο σεμινάριο που επικεντρώνεται προφανώς στις ε, προτάσεις για το άρθρο 85 και ένα ιδιαίτερα, το οποίο είναι το ότι η Eurojust, υπό του νέου κανόνε και κανονισμού, η Eurojust μπορεί να έχει εξουσίε και αρμοδιότητε να ξεκινά ερευνητικέ δραστηριότητε και να ξεκινά και διοκτικέ ε, δράσει. Είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Σαφώ υπάρχει περιθώριο για συζήτηση. Τι σημαίνουν όλα αυτά να ξεκινήσουν τέτοιε δράσει, δηλαδή ερευνητικέ δραστηριότητε. Σημαίνει μήπω ότι η Eurojust θα εκδίδει μια μη δεσμευτική σύσταση, μήπω θα σημαίνει ότι θα εκδίδει μια δέσμευση πρακτική σύσταση όσον αφορά ερευνητικέ δραστηριότητες, ανακρίσεις κτλ. Θα έχουμε λοιπόν ερευνητέ σε σχέση με τη Eurojust που θα ε, δίνουν συνέχεια σε τέτοιο είδους ε, δυνατότητες. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα τα οποία εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Όπως φυσικά εξετάζουμε και το θέμα για το άρθρο, υπό το άρθρο 86. Αν και πώς και με ποια δυνατότητα η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία θα μπορούσε να δημιουργηθεί, να συσταθεί όπως λέει και η συνθήκη. Πάλι εδώ υπάρχει περιθώριο για τη συζήτηση από τη Eurojust όσον αφορά αυτές τις δυνατότητες. Και αν επιτρέπετε θα ήθελα να, να στραφώ και να ολοκληρώσω λέγοντας, σας ευχαριστώ για την επισήμανση, στρεφόμενο στο θέμα της αξιολόγησης αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά την δημοκρατική λογοδοσία είναι ένα μια άλλη πτυχή που εξετάστηκε στο σεμινάριο της Μπρούις που προανέφερα. Και νομίζω σωστό είναι να πει κανεί ότι υπάρχουν <clears throat> διαφορετικές ε, πτυχές και θέματα σε σχέση με αυτό το εγχείρημα αξιολόγησης. Όλοι γνωρίζουμε φυσικά τις διατάξεις στη συνθήκη που απαιτούν να υπάρχει κοινοβουλευτικό έλεγχο, εποπτεία των δραστηριοτήτων τη Eurojust. Εντάξει, εδώ λοιπόν θα ήθελα να αναφέρω μόνο ίσω δύο γενικέ αρχέ ή προτάσει μάλλον περισσότερο που θα άξιζαν ίσω να εξεταστούν περαιτέρω και οι οποίε απορρέουν από αυτό το ε, σεμινάριο που έγινε πριν από δύο εβδομάδες στην Bruges. Πρώτα απ' όλα και υπό γενικού Μπορεί κανείς να πει, συνεχίζοντας τη συζήτηση που έλαβε χώρα και ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό, εχθές κιόλα, ότι υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ λογοδοσίας και ελέγχου όσον αφορά τις δραστηριότητες ενός οργανισμού σαν την Eurojust. Σίγουρα. Έχουμε λοιπόν στη Eurojust και έχουμε εμφανιστεί και συμμετάσχει με πολλές αφορμές ε, και ε, ενάψματα ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ΛΥΜΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι μια συνεισφορά αν θέλετε στην, στο εγχείρημα λογοδοσίας ε, της Eurojust ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν λοιπόν πιστεύω σε σχέση με αυτή την αρχή δεδομένη τη διαφορά μεταξύ ελέγχου και λογοδοσία, αν δεχθούμε αυτή τη διαφορά, απορρέουν διάφορα ερωτήματα. Θα, υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση για τη Eurojust και να βλέπει κανείς πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια από πλευρά της και έτσι να σταθμίζουμε και να μετράμε με τον αριθμό περιπτώσεων, για παράδειγμα, ή συσχετίζοντας και αξιολογώντας το πώς η Eurojust συνεισφέρει στο να βελτιωθεί η δικαστική συνεργασία. Θα έπρεπε κιόλας και αυτό είναι και ένα άλλο θέμα το οποίο εξετάστηκε στην πρωι. Θα έπρεπε η αξιολόγηση της Eurojust να συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση των συνεισφορών και παρεμβάσεων των κρατών μελών στο έργο της Eurojust. Διότι εδώ σαφώς η Eurojust μπορεί να προσθέσει πρόσθετη αξία, όπως προανέφερα, αν παίρνουμε από τα κράτη-μέλη επαρκή πληροφοριακά στοιχεία, επαρκείς πληροφορίες, έγκαιρα κιόλα. Αυτά είναι λοιπόν κάποια από τα στοιχεία που δημιουργούν ερωτήματα, κάποια από τα ερωτήματα τα οποία θίγονται και πρέπει να καλυφθούν ήταν αποτέλεσμα αυτή τη αξιολόγησης και του εγχειρήματο λογοδοσία. Έχω συνειδητοποιήσει ότι ξεπερνώ τον χρόνο μου και θέλω να προσθέσω αμέσως μια δεύτερη πρόταση που απορρέει από τις αρχικές συζητήσεις. Είναι πολύ πρώιμες ίσως σε πρώτη φάση συζητήσεις πώς θα έπρεπε να γίνει η λογοδοσία και τι πρέπει να γίνεται και με την αξιολόγηση. Με κάθε σεβασμό θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να εξεταστεί μια streamlined evaluation, δηλαδή μια εντεταγμένη σε αδρές γραμμές ε, ως εγχείρημα αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μας από πλευρά, της, από πλευρά σας και για αυτή την συνάντηση της ε, κοινοβουλευτική Επιτροπής σας ε, είχε ζητηθεί πριν από μια εβδομάδα να παρακολουθήσουμε μια συνάντηση από πλευρά της ε, Ισπανικής κοινοβουλευτική Επιτροπής μια και έχουμε 27 κοινοβούλια στα κράτη-μέλη 27 κράτη-μέλη και έχουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ΚΟΖΑΚ θα θέλαμε παρακαλώ να λάβετε υπόψη το φόρτο εργασίας και με ένα απλούστερο τρόπο σε αθρές γραμμές να μπορούν να γίνουν γίνονται όλα αυτά σε σχέση με εμά και εσά. Και σαν αποτέλεσμα όλων των συζητήσεων που είχαμε όσον αφορά την Eurojust, το αποτέλεσμα είναι ότι θέλουμε να συνεισφέρουμε στην αξιολόγηση και στις δραστηριότητες αξιολόγησης. Ελπίζουμε ότι κάτι μπορεί να προσθεθεί όσον αφορά την πείρα που έχουμε συλλέξει με τόσες ε, περιπτώσεις συνεργασίας που έχουμε με τις διοκτικές αρχές και τις εισαγγελίες. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Williams και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση των χρονικών ορίων που πρέπει να είναι σεβαστά. Και έχουμε και τους άλλους δύο εδώ στο πάνελ που παρακαλώ να και εκείνοι να προσπαθήσουν να τηρήσουν το χρόνο τους το πολύ 10 λεπτά ο καθένας ώστε να επαρκέσει ο χρόνος στις παρουσιάσεις τους και να έχουμε χρόνο για συζήτηση. Η κυρία Βέμπερ λοιπόν, εξ ονόματος της Επιτροπής ΛΥΜΕ, Πολιτικών Ελευθεριών της Ευρωβουλίας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχήν να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Williams για την παρουσίασή του. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω τη δυνατότητα ως εισηγήτρια του Κοινοβουλίου για τη Eurojust να μοιραστώ μαζί σας κάποιες από τις απόψεις μου για την πολύ σημαντική αυτή υπηρεσία. Είναι αλήθεια ότι έχουμε κάνει πολλά ε, ε, ειδικά ε, δεδομένου του γεγονότος ότι η υπηρεσία αυτή ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία. Έχουν γίνει πολλά και έχουν επιτευχθεί πολλά στο διάστημα αυτό, ο ε, κύριος Βίλιαμς ανέφερε την ε, αύξηση των ε, υποθέσεων, η οποία είναι εντυπωσιακή. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα πρέπει να πούμε ότι πιο συχνά τώρα τα κράτη-μέλη φαίνεται να αντιλαμβάνονται την αξία της ε, υπηρεσίας και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το συντονισμό ταυτόχρονων ερευνών αλλά και όσον αφορά την Συμφωνία Επικοινών Στρατηγικών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Αυτό φαίνεται και στην αύξηση του αριθμού των ε, συντονιστικών ε, ε, συναντήσεων. Αλλά τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει μόνο στην πράξη από τότε που ιδρύθηκε η Eurojust και σε θεσμικό επίπεδο έχουν γίνει πολλά. Πριν από λιγότερο από δύο χρόνια, το Δεκέμβριο του 2008, τροποποιήθηκε η ιδρυτική απόφαση της Eurojust για δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά που έγινε αυτό ήταν το 2003. και είμαι σίγουρη ότι στο μέλλον θα γίνουν και άλλες τροποποιήσεις διότι με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας ο ρόλος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων έχει αλλάξει σημαντικά. Το άρθρο 85 της συνθήκης αναφέρει σαφώς ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με κανονισμούς που έχουν υιοθετηθεί ε, με την κανονική νομοθετική διαδικασία θα ε, καθορίζουν την ε, δομή, τη επιχειρήση το πεδίο δράσης και τα καθήκοντα της Eurojust. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν είναι συνομοθέτης όσον αφορά την Eurojust. Και και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχουν στην ε, αξιολόγηση των ε, δραστηριοτήτων της Eurojust ε, σύμφωνα με την διάταξη αυτή. Τι σημαίνει αυτό, τι θα αλλάξει για την ίδια τη Eurojust. Εμείς σε τι ρόλο θα παίξουμε ως κοινοβούλια και πώς θα συνεργαστούμε μεταξύ μας. Και άλλες ερωτήσεις μου έρχονται στο νου. Δεν έχω απαντήσεις ακόμα αλλά πιστεύω ότι η συνάντηση αυτή αποτελεί καλή ευκαιρία να συζητήσουμε τα ερωτήματα αυτά και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε στη συνάντηση που έγινε πριν δύο εβδομάδες ε, από την... και οργανώθηκε από τη Βελγική Προεδρία. Δυστυχώς ε, οργανώθηκε κατά τη διάρκεια της ε, Συνόδου του Στρασβούργου. Ήμασταν υποχρεωμένοι να είμαστε παρόντες στην Ολομέλεια και αυτό ήταν κρίμα, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε συζητήθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα. Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε κάποιες ε, πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη εκεί και ε, αναρωτιέμαι μήπως μπορούμε να λάβουμε ε, ένα πιο αναλυτικό έγγραφο για τις συζητήσεις και τις προτάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής. Να επανέλθουμε στο σήμερα. Για να δούμε στην πράξη τι, ε, ποιοι θα είναι οι νέοι μα ρόλοι στη Eurojust θα πρέπει να περιμένουμε την πρόταση τη Κομισιόν. Τι μπορούμε να περιμένουμε όμω. Στο πρόγραμμα Στοχόλμη που υιοθετήθηκε πέρσι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε τα εξή. Ε, στον τομέα τη δικαστική συνεργασία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη τα κράτη-μέλη και η Eurojust να εφαρμόσουν πλήρω ε, την απόφαση του Συμβουλίου 2009 426 για την ενίσχυση της Eurojust που μαζί με την συνθήκη της Λισαβόνας παρέχει ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη της Eurojust τα επόμενα χρόνια συμπεριλαμβανομένης συμπεριλαμβανομένου των ερευνών που έχουν να κάνουν με την σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Με βάση την αξιολόγηση για την εφαρμογή του μέσου αυτού θα πρέπει να εξεταστούν σε δυνατότητες σύμφωνα με τις ε, σχετικές διατάξεις ε, της ε, συνθήκης συμπεριλαμβάνουν των νέων αρμοδιοτήτων που δίνονται στα εθνικά μέλη της Eurojust, την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του σώματος της Eurojust και τη δημιουργία ενός Ευρωπαίου εισαγγελέα. Σε, απάντηση σε αυτά η Κομισιόν ε, υιοθέτησε ένα, εκπώνησε ένα σχέδιο δράσης εφαρμογής του προγράμματος της Στοκχόλμης. Ε, προβλέπεται η ε, αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Eurojust το 2011 ενώ πρόταση κανονισμού που να δίνει στη Eurojust αρμοδιότητες να ξεκινάει έρευνας που κάνει έτσι πιο αποτελεσματική την εσωτερική δομή τη Eurojust και που, ε, όπου θα συμμετέχουν τα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλια και, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα υποβληθεί το 2012. Όπως όμως είπαμε νωρίτερα, η τελευταία τροποποίηση έγινε το 2008 ε, και το Κοινοβούλιο εξέφρασε την γνώμη του σε ε, νομοθετικό ψήφισμα το οποίο υιοθετήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του έτους αυτού. Ήδη τότε, όταν δεν ήταν ακόμα βέβαια η μοίρα της συνθήκης τη Λισαβόνα, ε, τονίσαμε την ανάγκη για αυξημένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ε, διασφαλιστεί ο ο καλύτερος δημοκρατικός έλεγχος. Ε, τότε δεν υπήρχε καμία υποχρέωση να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε όμως ε, το κοινοτικό δίκαιο εμπόδιζε το κοινοβούλιο από το να παίξει ε, ενεργό ρόλο στην εποπτεία των δραστηριοτήτων της Eurojust. Δυστυχώς καμία από τις προτάσεις μας αυτές δεν υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο. Μέχρι τώρα λοιπόν η επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι περιορισμένη. Ενημερωνόμαστε σχετικά με τις δουλειές που γίνονται από τη Eurojust με την ετήσια έκθεση, σχετικά με την έκθεση αξιολόγηση, σχετικά με την έκθεση της Κομισιόν ε, για την ε, εφαρμογή στα κράτη-μέλη, καθώς ε, και την έκθεση για τις δραστηριότητες των δικαστών συνδέσμων. Μόνο από το 2012 λοιπόν θα μπορέσουμε ε, να χρησιμοποιήσουμε τις νέες μας αρμοδιότητες και να συνηθίσουμε στους νέους, το νέο μας ρόλο ως ε, βουλευτές. Αυτό βέβαια δεν μας εμποδίζει από το να είμαστε προδραστικοί ήδη τώρα. Θα πρέπει να εκφράσουμε τις απόψεις μας, να συζητήσουμε μεταξύ μας σε πώς μπορούμε να ε, διαμορφώσουμε αυτή την ε, δημοκρατική λογοδοσία της Eurojust και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η λογοδοσία είναι το θέμα, δεν είναι ο έλεγχος των δραστηριοτήτων το θέμα. Ειδικά θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό δεδομένου ότι η παρούσα διατύπωση της συνθήκης ε, αφήνει σημαντικό περιθώριο ερμηνείας. Το άρθρο 85 και πάλι επαναλαμβάνω λέει ότι οι διατάξει αυτές θα πρέπει να ρυθμίζουν ε, ε, την συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της Eurojust. Έχουμε λοιπόν κάποιες σχετικές ερωτήσεις. Τι είναι οι δραστηριότητες της Eurojust? Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε Eurojust, εννοούμε το σώμα στο σύνολό του ή τα εθνικά μέλη. Θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό λοιπόν και κατά διάρκεια της σημερινής συζήτησης. Είμαι πεπισμένη ότι θα πρέπει να ανταλλάσσετε εμπειρίες και βέλτισες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο που εθνικά, εθνικοί φορείς ε, υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο και εποπτεία στα κράτη-μέλη. Η καλή συνεργασία είναι υψή τη σημασία για να μπορέσουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Προτού να κλείσω, να σχολιάσω σύντομα τι προβλεπόμενε ε, τροποποίησει ε, στην Eurojust, ιδιαίτερα τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τη και την ιδέα δημιουργία Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα. Όσον αφορά τη διεύρυνση των ε, καθηκόντων με την σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, η δυνατότητα της Eurojust να ξεκινάει ποινικέ έρευνες ε, ε, συμπεριλαμβάνεται κάτι που ανέφερε και ο Πρόεδρος. Να σας πω όμως ότι παρότι προτιμώ να ξεκινάω από τη θετική πλευρά, είμαι μάλλον επιφυλακτική σχετικά με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα όχι επειδή εγώ είμαι κατά της διεύρυνση των καθηκόντων, των αντίων, αλλά περιμένω να δω κατά πόσο θα συμφωνήσει το Συμβούλιο. Παρότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος Στοχόλμης, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η τελευταία αναθεώρηση της απόφασης Eurojust ε, μας ε, δίνει ε, σχετικές αποδείξεις. Δεν είμαι αφελής ώστε να πιστεύω ότι αυτό που εμεί θεωρούμε ότι θα είναι προ όφελο των πολιτών μας ε, γίνεται έτσι αντιληπτό και από τα κράτη-μέλη. Για αρκετού λόγου συμβαίνει αυτό. Καταρχήν το νομικό επάγγελμα είναι αρκετά συντηρητικό σε όλα τα κράτη-μέλη και ο συντηρητισμό αυτό αντικατοπτρίζεται ε, στον τρόπο που νομοθετεί το Συμβούλιο. Άλλο πολύ σημαντικό λόγο ε, έχει να κάνει με την προστασία των ε, αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη δεν βιάζονται να ε, μεταφέρουν τις ε, αρμοδιότητες αυτές σε ευρωπαϊκό φορέα. Και εδώ βλέπουμε ένα παράδοξο. Ενώ τα, οι ευρωβουλευτές είναι διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουν το σοβαρό έγκλημα, το διασυνοριακό έγκλημα, δίνοντα περισσότερε αρμοδιότητε στη Europol και στη Eurojust, τονίζοντα και την ανάγκη για πιο στενή συνεργασία επειδή η βασική μας ανησυχία είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία των δεδομένων, η πρόσβαση σε δίκες ε, δικαστικές διαδικασίες, ε, τα κράτη-μέλη άλλα λένε και άλλα κάνουν όταν νομοθετούν. Και πρέπει να πούμε ότι είναι δύσκολο για μας να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες μας πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης αν τα κράτη-μέλη τα ίδια δεν εμπιστεύονται τους ευρωπαϊκούς φορείς. Επιτρέψτε μου να πω και λίγα για τη δημιουργία Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Η δυνατότητα προβλέπεται στην συνθήκη, ε, όταν όμως κοιτάμε την πραγματικότητα, μάλλον μοιάζει με αυταπάτη αυτό προς το παρόν. Αυτή τη στιγμή νομίζω θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ε, ενίσχυση της Eurojust και των δραστηριοτήτων τας, ε, να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των κρατών μελών στις έρευνες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως και να έχει, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι γνώμες των Ευρωπαίων πολιτών και σκέφτομαι ιδιαίτερα δύο μέσα, την άμεση επικοινωνία και δεύτερον μέσω τέτοιων συναντήσεων με μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, διότι εσείς εκπροσωπείτε τους Ευρωπαίους πολίτες στα εθνικά σας κοινοβούλια. Ελπίζω η συνάντηση αυτή να είναι το ξεκίνημα μιας μακράς και επικοδομητικής συνεργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Βέμπερ. Έτσι θα είναι όπως είπατε. Και τώρα η κυρία Κριστίν Τεφέν από την Βελγική Γερουσία. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γαλλικά. Πολλά καλύφθηκαν ήδη από τους συναδέλφους σήμερα το πρωί. Όμως το πώς λειτουργεί η Eurojust το είδαμε ήδη από κάποιες μαρτυρίες. Επιτρέψτε μου τώρα να έρθω στο πλαίσιο, στο σκηνικό, εντός του οποίου γεννήθηκε η Eurojust. Διότι δεν είναι ότι δεν γνωρίζετε την ιστορία εντός του οποίου έγινε αυτή η γέννηση, αλλά υπάρχουν ακόμη κάποιες δυσκολίες επί της πράξης και θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα, τις δυσκολίες που θα πρέπει να διορθωθούν και να αντιμετωπιστούν. Ίσως η Eurojust ασχολείται εδώ με προνόμια που τα κράτη-μέλη θεωρούν ε, πολύ δικά του και πολύ προσφυλή ακριβώ επειδή έχουν να κάνουν με την ε, έννοια της αυτοκυριαρχίας τους την ίδια. Και δεν είναι απλό να παραδώσουν αυτά τα προνόμια. Άλλωστε και το δικαίωμα πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή σε θέματα ποινική δικαιοσύνη ήταν, περιορισμένα, ήταν περιορισμένες και ήταν ένα θέμα των εθνικών κυβερνήσεων και η συνθήκη του Άμστερνταμ έδωσε και τη γέννηση, έδωσε δικαίωμα στο Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο να γεννηθεί με ένα ευρύτερο εγχείρημα. Ένα εγχείρημα θεωρητικό με κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Ένα εγχείρημα λοιπόν, ένα σχέδιο αλλά και με κάποιο πρακτικό σκέλος. Τώρα το σύστημα αυτό ποινική δικαιοσύνη, ε, προκειμένου να επιτρέψει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, έχει καθυστερήσει σε σχέση με το σύστημα αστυνομική συνεργασία. Ένα σύστημα που δημιουργήθηκε πολύ πιο γρήγορα. Ακριβώ γιατί η Europol αρχίζει να λειτουργεί από το 1995 με την ε, πρώτη δημιουργία του χώρου του Σέγγεν. Το σύστημα λοιπόν, το, το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχικά βασίστηκε σε ελάχιστα στοιχεία. Γιατί υπήρχε μια σχέση διαλεκτική μεταξύ των όσων υποστήριζαν μια διακυβερνητική προσέγγιση, αρκετά αυστηρή, και όσων ήθελαν μια υπερεθνική προσέγγιση. Θα θυμάστε την απόφαση τη συνεδρίαση μάλλον δικαστών των Ευρωπαϊκών χωρών στη Γενέβη το 1996, οι οποίοι ε, εξέφρασαν ε, την διαμαρτυρία τους για το ότι η διασυνοριακή εγκληματικότητα θυμίζει το σύννεφο διενεργό του Τσερνομπίλ. Δεν σταματάει στα σύνορα, τα ξεπερνάει και βεβαίως αυτό θα πρέπει να απασχολήσει και το δικαστικό σύστημα. Άλλωστε και στο νομικό σύστημα υπάρχουν απόψει και υποστηρικτέ όπω κυρία Ντέλμα που έχει προτείνει κανόνε ε, ε, προκειμένου να προστατευτούν τα οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κανόνε που είναι σύμφυτοι με την δημιουργία τη Ένωση. Γιατί πραγματικά η οικονομική εγκληματικότητα δεν σταματάει στα σύνορα. Ήδη στο Τάμπερ ε, το 1999 ακούσαμε λοιπόν τι πρώτε ιδέε για το θέμα αυτό και κάπω επώδυνα τα κράτη-μέλη κατάλαβαν ότι πρέπει να δώσουν μια διαθεσμική απόκριση στι ανάγκε αυτέ, μια συστημική απάντηση. Αυτό ήρθε και ω λογική συνέπεια μεταξύ την δημιουργία των δικαστών συνδέσμων το 1996 και το δικαστικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1998. Όμως αυτά όλα σε βάση πειραματική, δοκιμαστική και ω μια προσωρινής υπηρεσίας που δεν είχε ακόμα τη μορφή της Eurojust. Όμως η απόφαση του Συμβουλίου τη 28 Φεβρουαρίου 2002 έδωσε, έτρεψε στη Eurojust να κάνει τα πρώτα της βήματα. Στο Βέλγιο τώρα ξέραμε μια ενδιάμεση, γνωρίζαμε μια ενδιάμεση λύση, μια, μια δομή συνεργασίας και συντονισμού όπου για τους υπέρμαχους ε, της διακυβερνητικής προσέγγισης δεν ε, εμπλέκεται με τις ε, κρατικές πρωτοβουλίε και τα κρατικά προνόμια. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικαστικού Σώματο. Συζητήθηκε στην Επιτροπή Δικαιοσύνη το θέμα αυτό, στη Βελγική Γερουσία, προκειμένου να καθορίσουμε το ανάλογο πλαίσιο και οι εθνικοί βουλευτές εξέφρασαν την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει σαφώς δημοκρατικός έλεγχος σε ένα τέτοιο σύστημα, ενώ πολλοί γερουσιαστές σχολίασαν την απουσία διαφάνειας και προβολής των αποφάσεων πλαίσιο οι οποίε θα πρέπει και αυτέ να υπόκεινται σε δημοκρατικό έλεγχο. σω το είδο τη συζήτηση που έχουμε σήμερα να μπορέσει να αντισταθμίσει αυτή την έλλειψη. Και είναι ένα βήμα προ την σωστή κατεύθυνση. Ίσως τα εθνικά κοινοβούλια αποδείξουν ότι δεν ε, εκφράσαμε απόψεις ε, στο κενό και ότι θα μπορέσουμε να επιτελέσουμε πρόοδο. Έτσι λοιπόν για τη Eurojust, αφού είδαμε το παρελθόν της, ας δούμε τις προοπτικές της. Το 2009 πλέον είδαμε ότι οι υποθέσεις που εξέτασε η υπηρεσία συνεχώς αυξάνονται. 15% παραπάνω το 2008 με 2009. Σημαίνει αυτό άραγε ότι υπάρχουν περισσότερες υποθέσεις, περισσότερες περιπτώσεις, περισσότερες παραβάσεις ή ατασταλίες ή σημαίνει ίσως ότι συλλέγονται με πιο ακριβή τρόπο, πιο προσεκτικό τρόπο τα δεδομένα, ότι είναι πιο αποτελεσματική η δίωξη την αύξηση των αριθμών των στατιστικών στοιχείων δεν πρέπει να συμπεράνουμε ότι υπάρχει απαραίτητα και αύξηση της διασυνοριακής ε, εγκληματικότητας. Απλώς είναι καλύτερα γνωστή η δραστηριότητα της Eurojust και καλύπτει επίσης η ίδια καλύτερα τις ε, πρακτικές ανάγκες. Ποιε είναι τώρα οι προκλήσεις που προκύπτουν. Η συνθήκη της Λισαβόνας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα σώμα ε, εισαγγελέων ευρωπαϊκό. Είναι αλήθεια ότι η δημιουργία ενός τέτοιου σώματος βάσει της Eurojust θα άλλαζε ε, σημαντικά την προοπτική, το πλαίσιο και την εικόνα. Η εικόνα αλλάζει πολύ για την άσκηση των δραστηριοτήτων της Eurojust. Μπορεί όμως ένα τέτοιο σώμα να λύσει όλα τα προβλήματα. Στην αρχή της παρουσίασής μου μίλησα για το πώς ε, ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να ε, συνδυαστεί με την αρχή της διακυβερνητικής λειτουργικότητας και την κυριαρχία των κρατών. Ένα τέτοιο λοιπόν σώμα είναι τόσο αναγκαίο ότι είναι, δεν αφισβητεί τόσο πολύ, αλλά θα είναι και αποτελεσματικό διότι η δημιουργία ενό σώματο αγγελών στην Ευρώπη θα σημαίνει ότι το να έχουμε τις δυνατότητες δίωξης δεν μας οδηγεί και στην δυνατότητα κίνησης ε, ποινικών νομικών ε, διαδικασιών. Δηλαδή τα πάντα θα εξαρτηθούν από τους κανόνες που θα διέπουν ένα τέτοιο σώμα. Βεβαίως, συνολικά μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι ατασταλείς παρανομίες οι οποίες κάποια στιγμή εκδικάζονται, είναι περίπου ίδιε ε, στα περισσότερα κατημέλη. Όμω δεν είναι βέβαιο ότι αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό πρέπει να το δούμε. Δημιουργία λοιπόν σώματο εισαγγελέων στην Ευρώπη, ναι, αλλά με τι μορφή. Διότι πρέπει να δούμε τι νομική πολιτική θα ασκηθεί από αυτό το σώμα. Και αυτό το σώμα επίση ε, ενώπιον ποιου θα λογοδοτεί. Ε, από την άλλη, αν υπάρχει ένα οργανισμό δίωξη ευρωπαϊκό, τίθεται και το εξή ερώτημα που σχετίζεται με τι προκλήσει που θα πρέπει να απαντήσουμε στο μέλλον. Ποιο τελικά θα εφαρμόζει του κανόνε. Τελικά ποιο θα αποδίδει δικαιοσύνη, διότι δεν φτάνει να εκδικάζονται οι υποθέσει. Πρέπει τελικά να φτάνουν και σε αίσιο πέρα όλε αυτέ οι προσπάθειε, δηλαδή να δικάζονται οι εγκληματίε και να αποδίδεται δικαιοσύνη. Τα κατοπινά δηλαδή στάδια, η συνέχεια τη διαδικασία. Ξέρουμε ότι το τομέα τη ευρωπαϊκή ποινική δικαιοσύνη βρίσκεται στα πρώτα του βήματα. Ίσως προχωρά ψελίζοντας ε, και με ασταθές βήμα. Όμως στο άμεσο μέλλον πρέπει να δημιουργηθούν προφανώς κοινοί κανόνες, αλλά και μια πραγματική ποινική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι τι διάρθρωση θα υπάρχει, τι θέση θα καταλάβει η Eurojust μεταξύ όλων αυτών των φορέων, εάν δεν έχει ήδη καταρτιστεί η Ευρωπαϊκή Ποινική Πολιτική. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις απόψεις σχετικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ντεφρέν. Και τώρα έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε. Θα ακούσουμε τους συναδέλφους. Έχουμε ένα σύντομο κατάλογο αγορητών και θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους που θα παρέμβουν να περιοριστούν σε δύο λεπτά παρέμβασης ώστε να έχουμε όλοι το χρόνο να μιλήσουμε και να έχουμε και τις απαντήσεις των ε, συμμετεχόντων. Ο κύριο Σαϊχουμπέρο από την Ισπανική Βουλή. Πολύ σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Χων Φερνάντο, θέλω να ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον και αυτών των κοινοβουλευτικών ημερίδων και να πω ότι με αυτέ τι ημερίδε επίση υλοποιούμε αυτό το οποίο προβλέπεται από τη συνθήκη τη Λισαβόνα, το άρθρο 85, συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων τη Eurojust ο ίδιο ο κύριο Βίλιαμ, ο οποίο ανέφερε αυτό το θέμα και θέλω να τον συγχαρώ διότι για πρώτη φορά ήρθε στη δική μα μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή στις, στη Βουλή μα για να, μπορέσει, να, να μπορέσουμε να συζητήσουμε με του κοινοβουλευτικού εκπροσώπους και του γερουσιαστέ για το τι γίνεται από πλευρά Eurojust. Εμεί θεωρούμε ότι μια φορά ετήσια θα ήταν αναγκαία αυτή η παρουσία. Το ανέφερε και ο κύριος Βίλιαμ και του χρόνου θα έχουμε και προηγούμενα ερωτήματα τα οποία θα έχουν ε, διατυπωθεί για να εξεταστεί καλύτερα τι γίνεται με τη Eurojust. Γι' αυτό με οδηγεί στο να θέσω επιτραπέζι στην ανάγκη να υπάρξει μια κοινή διαδικασία αξιολόγηση ε, όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια για αυτέ τι δραστηριότητε και στι επόμενε δραστηριότητε μα στην ΚΟΣΑΚ ε, να μπορέσει να διατυπωθεί ο ρόλο σε σχέση με την Eurojust εκφράζουμε ικανοποίηση για τις ε, προόδους που έχουν σημειωθεί όσον αφορά την πάροδο των ετών με τη λειτουργία της Eurojust και για τις προσπάθειες που κάνουν τα εθνικά κοινοβούλια από πλευρά τους για να προσαρμόσουν το ποινικό δίκαιο και το δικονομικό πλαίσιο μέσα στις νέες αυτές εξελίξεις για την αντιμετώπιση αυτών των ε, περιπτώσεων που αφορούν την Ένωση. Θα ήθελα να κάνω αναφορά και έγινε αυτό σε σχέση με την Προεδρία, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υποστηρίζουμε τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία των συμφερόντων, δημοσιονομικών, οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και η κυρία Ντεφρένια που είναι παρούσα εδώ θα πρέπει να δούμε ποιες αρμοδιότητες θα έχει αυτή η Γενική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και μέσα σε δύο δευτερόλεπτα να μπορούσαμε να δούμε αν μπορεί να υπάρξει κάποιο σχόλιο από την Προεδρία. Ποια είναι η αξιολόγηση σε σχέση με τις κοινέ ομάδες έρευνας από τη Eurojust, κοινέ ερευνητικές ομάδες και ποια είναι ακόμα και τα αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων δικαιοδοσίας σε σχέση με την Eurojust. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μαριτάτη από την Ιταλική Γερουσία, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας, που βρίσκω ότι πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο, ίσως και για πρώτη φορά. Η συμβολή μας, λοιπόν, ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμη. Επικροτώ λοιπόν τι αλλαγέ που επισυμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Eurojust από τότε που γεννήθηκε ο οργανισμό. Βεβαίω έχει ακολουθήσει σωστή κατεύθυνση το ίδιο και η Ευρώπη διότι πλέον μιλάμε για περιεχόμενο και δομέ που μπορούν να δώσουν στον οργανισμό αυτό μια συγκεκριμένη λειτουργία και ένα νόημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Θα πρέπει όμω να είμαστε σαφεί και να μην προτρέχουμε διότι η συνθήκη τη Λισαβόνα ε, προβλέπει συγκεκριμένο περιεχόμενο και αρμοδιότητε ώστε να ξεκινήσουμε και ποινικέ διαδικασίε. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να αποσαφηνίσουμε το εξή. Στην Ιταλία έχουμε μακρά εμπειρία που θα μπορούσε να διευκολύνει τον ε, προγραμματισμό μα εδώ, λόγω των δράσεών μα κατά τη μαφία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με το εισαγγελικό σώμα το εθνικό, που αρχικά ε, για κάποια εγκλήματα λειτουργεί ως, ε, σε εθνικό επίπεδο. Όμως κάποιες φορές εκεί είχαμε και σοβαρέ αντιστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε αυστηροί και σκληροί και σε εθνικό επίπεδο. Θα ήταν λοιπόν σφάλμα κατά την άποψή μου, θα ήταν επικίνδυνο να θα προβλέψουμε όλα αυτά τώρα, να, θα προτρέχαμε εάν η Eurojust ε, υποκαταστήσει ένα ευρωπαϊκό εισαγγελικό σώμα που θα μπορούσαν με τη σειρά τους να υποκαταστήσουν τα εθνικά εισαγγελικά σώματα ή να αναλάβουν κάποιες από τις λειτουργίες τους. Η Eurojust και το εισαγγελικό σώμα της Ευρώπης δεν μπορεί να, θα μπορούσαν να έχουν ανάλογες δραστηριότητες με το εθνικό μας ε, σώμα κατά της μαφίας, δηλαδή γνώσεις και πληροφορίες μέσω της υποχρεωτικής εφαρμογής εφαρμογή και συλλογή δεδομένων που κάποια, τα κάτι μέλη θα πρέπει να συλλέγουν και να παρέχουν μέσω των εθνικών του ερευνών. Ο συντονισμό λοιπόν, συντονισμό που προβλέπει και συνδρομή, είναι θετικό βήμα ε, και να υπάρχει και υποκίνηση. Να προβλέπεται όμως μην δραστηριότητα που να υποκαθιστά την εθνική δράση είναι κάτι πολύ πρόημο και αδικαιολόγητο. Το πλαίσιο λοιπόν της Eurojust που να συνδέεται με ένα ευρωπαϊκό εισαγγελικό σώμα είναι μια σωστή ιδέα αλλά να μην θίξει τα προνόμια και την κυριαρχία των εθνικών κρατών μελών. Να συνοδεύει αυτές τις αρμοδιο... αυτήν την ε, εθνική κυριαρχία και τα... τη δυνατότητα πρωτοβουλίας. Αλλά η δράση η δίωξη μάλλον του διακρατικού εγκλήματος θα μπορούσε να υποβοηθηθεί από ένα τέτοιο σώμα. Ο έλεγχος της εγκληματικότητας, ο έλεγχος της νομιμότητας, της δράσης δεν μπορεί να εμπλέκεται με τα εθνικά όρια. Να έχει πολιτική ε, φύση, αλλά σε καμία περίπτωση να μην ε, παρεμβαίνει στα εθνικά. Ευχαριστούμε ο κύριος Ντιάς Ντεμέρα από την Επιτροπή Λίμπερ. Ευχαριστώ πρόεδρε πολύ σύντομα υπόρους ε, ρεαλισμού και για να προκαλέσω κάποια συζήτηση σε σχέση με τις ομάδε εργασίας στο σεμινάριο της Μπούζ. πιστεύω κύριε Πρόεδρε του σώματος ότι το Συμβούλιο θα συμφωνήσει με το να ξεκινήσουν οι δραστηριότητες, οι ερευνητικές δραστηριότητες. Βρισκόμαστε περισσότερο πια στην πορεία του να προταθούν ή να προταθεί η έναρξη αυτών των δραστηριοτήτων. Μεταξύ άλλων νομίζω σκόπιμο είναι να κάνουμε μια αποσαφήνιση όσον αφορά το τι εννοούμε με έλεγχο. Έλεγχος σημαίνει να γνωρίζει κανείς από πλευρά των πληροφοριών και να απαιτεί ευθύνες όχι μόνο πληροφορίες ή να παίρνει πληροφορίες αλλά να ζητεί να αποδοθούν ευθύνες. Και υπό το πλαίσιο του ρεαλισμού αυτή η αξιολόγηση και αυτή η λογοδότηση θα πρέπει να παιρνει πληροφοριες αλλα να ζητει να αποδοθουν ευθυνε και υπο το πλαισιο του επίσης τον όγκο πληροφοριών που παίρνει η Eurojust από τα κράτη-μέλη. Να ελέγχουμε είναι ένα ρήμα πολύ εύκολο που χρησιμοποιείται συχνά και το κατανοούν στα εθνικά κοινοβούλια. Έτσι αναλογικά με αυτό που κάνουν τα εθνικά κοινοβούλια έτσι εννοείται ο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Να απαιτεί κανεί ευθύνε με βάση τι πληροφορίε που έχουν στη διάθεσή του και να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να απαιτήσουν ευθύνε. Περισσότερο έλεγχο, περισσότερη εμπιστοσύνη. Λιγότερο έλεγχο, μεγαλύτερη θολότητα. Πιο θολό τοπίο. Και γι' αυτό σε σχέση με την εισαγγελία, τη Γενική Εισαγγελία, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρέπει να είμαστε πάλι ρεαλιστέ και συμμερίζομαι αυτό που είπε η Ρενάτε Βέμπερ. Και είναι αυτό που είχα πει και εγώ χθε. Αυτό είναι κάτι αυτή τη στιγμή που μοιάζει με μια χήμερα. Καμιά περιτροπή σε εναλλασσόμενη προεδρία δεν θέλει να μιλήσει γι' αυτό ή να δεσμευθεί. Και τέλει, εν τέλει, πρόεδρε, ένα ποινικό ευρωπαϊκό δίκαιο και αυτό είναι κάτι το ανέφικτο ή το αδύνατο αυτή τη στιγμή πιστεύω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Από πλευρά τη Βουλής ε, των Λόρδων, ε, παρακαλώ εσείς, ε, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση. Στην χθεσινή μα συζήτηση για την Europol εχθές υπέβαλα μια πρόταση και διατύπωσα ένα ερώτημα. Η πρόταση είναι η εξή. Τα άρθρα τα οποία συσχετίζονται με την κοινοβουλευτική ελεγκτική δραστηριότητα όσον αφορά τη συνθήκη τη Λισαβόνα έχουν διαφορετική διατύπωση για τη Europol και τη Eurojust. Είναι δύσκολο όμω να αξιολογήσει κανεί για ποιου λόγου υπάρχει αυτή η πρακτική διαφορά στι διατυπώσει σε αυτέ τι αντίστοιχε ρήτρε. Έτσι, οποιασδήποτε διαδικασίε αναπτυχθούν για την κοινοβουλευτική ελεγκτική δραστηριότητα θα πρέπει να είναι απλέ. Και δεν πιστεύω εγώ να υπάρχει οποιοδήποτε λόγο, γιατί αυτέ οι διαδικασίε θα έπρεπε να είναι διαφορετικέ για μια οργάνωση, για έναν οργανισμό σε σχέση με έναν άλλον. Αυτό σίγουρα θα είχε το όφελος να μας, εξοφ... μας εξοικονομήσει πολύ μεγάλο χρόνο και όσον αφορά και τις συζητήσεις αν είχαμε ένα κοινό πλαίσιο αυτών των διατάξεων και για τα δύο όργανα. Είναι κέρια σημασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια να δεχθούμε και να κατανοήσουμε ότι κάνουμε λόγο για λογοδοσία εδώ και όχι για έλεγχο. Και η ερώτησή μου εχθέ το απόγευμα ήταν και την ξαναδιατυπώνω σήμερα το πρωί και ελπίζω ότι εσεί, Πρόεδρε, εσεί θα διαβιβάσετε αυτή την πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντηθεί. Γιατί προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπάρχει κοινοβουλευτική εποπτεία για τη Eurojust το 2012 αλλά για το, μέχρι το 2013 δεν θα υπάρξει τέτοια για τη Europol. Τι μπορούμε να κάνουμε, να επισπεύσουμε αυτές τις ημερομηνίες, να τεθούν πιο νωρίς, διότι η λογοδοσία κοινοβουλευτική είναι τεράστια σημασία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τα Εθνικά Κοινοβούλια υπό το πρίσμα των διευρυμένων αρμοδιοτήτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο με τις συνθήκες Λισαβόνα. Λισαβόνας. Αν πάρουμε το χρόνο να απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις που εθίγησαν σήμερα το πρωί, θα μπορούσε ακόμα περαιτέρω να μετακινηθεί αυτή η ημερομηνία. Δεν έχει νόημα λοιπόν να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες ε, δημοκρατικής λογοδοσίας πιο νωρίς ε, πριν από οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σας ευχαριστώ. Ο κύριος Στενάλια από το, την Ιταλική Βουλή παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η συνθήκη της ε, Λισαβόνας άνοιξε νέους δρόμους ως προς το σύνολο κανόνων του ποινικού δικαίου και του αστικού δικαίου και σε σχέση με το δικαστικό σύστημα απαιτεί και συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων πολύ πιο έντονη. Για αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση είναι ιδιαίτερη σημασία, διότι είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα πρέπει λοιπόν η τάση αυτή να ενισχυθεί κατά την άποψή μου μέσω συγκεκριμένων δομών και με συγκεκριμένους τρόπους και μεθοδολογίες εργασίας. Κατά πρώτον, θα πρέπει να δούμε την ανάγκη για τέτοια ζητήματα, να υπάρχει μια προκαταρκτική διαβούλευση με τα εθνικά κοινοβούλια, ε, ώστε να αποφανθούν και όταν πρόκειται να καθοριστούν τα συστήματα λειτουργίας της Europol και της Eurojust. Θα πρέπει τέτοιου είδους συνεδριάσεις και συναντήσεις να γίνουν συστηματικές και συχνές, έχοντας υπόψη την ουσία της σημερινής συζήτησης. Πιστεύω ότι για την Eurojust ε, θα πρέπει όπως σωστά ήδη παρατηρήθηκε, να δούμε το πρόβλημα του ελέγχου ε, του ελέγχου στο σωστό επίπεδο. Δηλαδή άλλο θέμα είναι ο συντονισμό και άλλο δημοκρατικός έλεγχος για τη Eurojust. Ιδίως για τις ε, εξελίξεις που ο οργανισμός αυτός θα γνωρίσει χάρη στην εφα... λόγω της εφαρμογής μάλλον της συνθήκης της Λισαβόνας. Βέβαια τα βήματά μας θα πρέπει να είναι μικρά και διστακτικά. Αλλά το να αρχίσει η έρευνα, να ασκηθεί η ποινική ευθύνη, να συντονιστούν οι ποινικέ έρευνες του οργανισμού αυτού, ε, να επιληθούν οι διαφορές αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας, όλα αυτά ε, αφορούν πολύ ευαίσθητε πτυχές του προβληματισμού των κρατών μελών ω προς την υποχρεωτική εκτέλεση κάποιων ε, νομικών πράξεων λόγου χάρη που για μας ε, στη δική μας νομοθεσία είναι θέμα μέχρι και συνταγματικό. Έτσι λοιπόν απαιτείται από τη Eurojust για τις λειτουργίες τους, για τις λειτουργίες της αυτές, να καθορίσει κριτήρια προκαταρκτικής αποτίμησης και αξιολόγησης της δραστηριότητάς της. Τα κριτήρια αυτά θα αφορούν γενικότερα την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της και όχι την εξέταση επιμέρους υποθέσεων. Τώρα, το να υπάρχει ένα εισαγγελικό σώμα ευρωπαϊκό, αυτό απαιτεί ενισχυμένη συνεργασία. Και μια τέτοια ιδέα βάσει του ποινικού δικαίου θα πρέπει να... Ε, μια τέτοια ιδέα θα πρέπει να, είναι, να την αντιμετωπίσουμε με τρόπο πολύ συνετό. Γιατί πραγματικά μπορεί να υπάρχουν και πολύ σοβαρέ συνέπειε για τι εθνικέ νομοθεσίε. Ευχαριστούμε ο κύριο Μόλτερ από την Επιτροπή Λίμπερ. Yes. Thank you. Ευχαριστώ. Πριν πολύ καιρό ήμουν μέλος της πρώτης εξεταστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις απάτες ε, στο, στις περιπτώσεις transit. στα τέλη της δεκαετίας του 90, μια από τις σημαντικές συστάσεις ήταν να υπάρχει Ευρωπαίος εισαγγελέα. Μετά από τόσα χρόνια, διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατόν, δεν είναι εφικτό σε αυτό το πολιτικό κλίμα. Αυτό με εκπλήσει. Θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη της Eurojust σχετικά με την αναγκαιότητα ή όχι ε, αυτού του μέτρου. Προβλέπεται στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Μερικοί θεώρησαν ότι είναι μεγάλος τρίαμβος αυτό, ενώ τώρα μερικοί αντιδράνε. Είναι καλό αυτό ή κακό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζαβάρα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει μια αρχαία ελληνική ρίση, σύμφωνα με την οποία αποτελεί αρχή σοφίας των ονομάτων η επίσκεψη. Γι' αυτό θεωρώ ότι για να μην έχει τελετουργικό χαρακτήρα αυτού του είδους οι συναντήσεις, θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε πλήρως τι νόημα δίνουμε στις έννοιες του δημοκρατικού ελέγχου, της λογοδοσίας και της αξιολόγησης. Διαφορετικά θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να μιλάει με ωραίες ιδέες, αλλά η αποτελεσματικότητα αυτών των ιδεών να είναι μηδενική. Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι δεν μπορεί κανένας να μιλάει για μια προοπτική δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα εάν προηγουμένως δεν έχει εντάξει αυτό το θεσμό μέσα σε ένα σύστημα δικαιοδοτικής λειτουργίας της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν μαζί με τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα να είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε και για ένα Ευρωπαϊκό Ποινικό Δικαστήριο, για ένα σύστημα δηλαδή δικαιοδοτικό στον τομέα του ποινικού δικαίου. Διαφορετικά δεν θα έχει κανένα νόημα η οποιαδήποτε αναφορά και προοπτική. Μια τρίτη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι το πέρασμα από το σημερινό στάτους της, Eurojust σε εκείνο όπου θα μπορεί να έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα στα πλαίσια της ε, ε, μιας ποινική δικαιοδοσίας είναι το πέρασμα σε μια άλλη ποιότητα για την οποία θεωρώ ότι δεν υπάρχουν σήμερα ούτε πολιτικά ούτε κοινωνικά ούτε εθνικά οι προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση θέλω να πω και εγώ ότι είμαι μέλος της Επιτροπής του Ελληνικού Κοινοβουλίου που εξετάζει το σκάνδαλο Siemens. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω από πλευράς Eurojust για ένα τέτοιο διασυνοριακό έγκλημα στο οποίο έχει αποδειχθεί ότι έχουν διαφθαρεί κρατική και πολιτική λειτουργή στην Ελλάδα και έχει ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο σε δισεκατομμύρια ευρώ, ποια είναι η μέχρι σήμερα συνεισφορά της Eurojust και τελευταίο θα ήθελα να ξέρω γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε έτοιμοι σε αυτό το τομέα τουλάχιστον που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ίδρυση και τη συγκρότηση του ενιαίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης να ξέρουμε στον τομέα της δίωξης του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος που έχει σχέση με τη διαφθορά πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων ποια είναι τα μέχρι σήμερα στατιστικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Νομίζω ακούσαμε αρκετέ ενδιαφέρουσε παρατηρήσει. Βλέπω και άλλο συνάδελφο θέλει το λόγο, ο κύριο Ρόγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μπορούσαν οι αστυνομικέ δυνάμει των 100 μελών αντί να δαπανούν του πόρου του ε, για να ερευνούν και να κάνουν συλλήψει, να εκδίδουν εντάλματα για διακρατικά εγκλήματα που δεν έχουν διαπραχθεί στη δική τους επικράτεια. Δεν θα μπορούσαν αυτά λοιπόν να γίνουν αποτελεσματικότερα με συντονισμό. Διότι υπάρχουν θέματα λόγω χάρη ελευθερίας έκφρασης που μπορεί μέσω του διαδικτύου σε μια χώρα με περισσότερο αυστηρά συστήματα να ξεκινούν από άλλες χώρες. Κάτι που συνέβη πρόσφατα στις κάτω λόγω χάρη οι, τα επικριτικά σχόλια κατά του Ισλάμ θεωρούνται αδίκημα στην χώρα αυτή και όχι σε άλλες ας πούμε. Ο κυρία Ντεφρέν έδωσε εν μέρη μια απάντηση στο θέμα αυτό λέγοντας ότι θα πρέπει όλοι να έχουμε κοινούς νόμους. Αλλά αυτό θα πρέπει να μην ε, πλήττει καθόλου την εθνική κυριαρχία, όπω είπαμε. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Έχουμε τελικά λίγο χρόνο για απαντήσει από του ε, συμμετέχοντέ μα, του προσκεκλημένου μα. Θα του παρακαλέσω να είναι στο δυνατόν πιο σύντομοι. Κύριε Βίλιαμ. Um, um, uh, Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω δύο πράγματα να συναγάγω κυρίως από τις πολλές, ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις, ε, ερωτήσεις και σχόλια που έγιναν. Το πρώτο αφορά την λογοδοσία και τον έλεγχο. Πιστεύω ότι από ό,τι φαίνεται υπάρχει κάποια συνένεση όσον αφορά την σπουδαιότητα της λογοδοσίας υπό πραγματικούς όρους χωρίς να προσπαθεί κανείς να διασφαλίσει τον λειτουργικό έλεγχο, δηλαδή έλεγχο επί συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και περιπτώσεων. Και αξίζει να τονίσουμε σε αυτό το πρίσμα ότι ήδη στην Eurojust υπάρχουν εθνικοί εκπρόσωποι που συντάσσουν εκθέσεις και τις υποβάλλουν στις εθνικές τους αρχές και σε κάποιες περιπτώσεις επίσης και τις υποβάλλουν και στα εθνικά κοινοβούλια, στα εθνικά κοινοβουλευτικά σώματα και αυτό είναι κάποια ίσως ένδειξη πώς τα πράγματα θα μπορούσαν να εξελιχθούν και να συνεχιστούν στο μέλλον. Όμως ακόμα διατηρείται η διαφοροποίηση, η διαφορά μεταξύ λογοδοσίας και ελέγχου. Ταυτόχρονα όμως είναι ένα θέμα εταιρικότητας μεταξύ Eurojust και Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πώς αυτή η σχέση μπορεί να ενδυναμωθεί ακόμα περαιτέρω. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο απορρέει και το οποίο είναι αντικείμενο διαφορετικών παρεμβάσεων και αυτό. Αφορά αυτό το γραφείο του Ευρωπα... Ευρωπαίου Εισαγγελέα, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σημαντικό είναι να θυμόμαστε εδώ το ότι όσον αφορά την προοπτική στο παρελθόν και την εξέλιξη της Eurojust, ότι αυτό είναι ένα θέμα σαφώς το οποίο αφορά πολιτική λήψη απόφασης. Είναι καθαρά πολιτικό θέμα και δεν είναι θέμα απόφασης της Eurojust προφανώς. Αυτό όμως το οποίο μπορεί να κάνει η Eurojust όσον αφορά αυτή τη συζήτηση είναι να συνεισφέρει και ελπίζουμε με θετικό νόημα και πρίσμα για την συζήτηση αν θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό όργανο εισαγγελίας ή όχι με την πείρα που έχει η Eurojust με ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις και την ε, διαφώτισή τους. Όταν έχουμε περιπτώσεις που ε, μπλέκουν παραβιάσεις και παραβάσεις ε, των συμφερόντων, οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρεαλιστικό αυτό θα πρέπει να είναι το επίκεντρο θα έλεγα του, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αν δημιουργηθεί και ξεκινήσει τη λειτουργία του αυτό το όργανο. Σαφώς προβλήματα έρευνας και δίωξης ακολουθούν αμέσως στην ιεράρχηση, στην αλυσίδα και είναι σημαντικό να το δούμε αυτό για την Eurojust στο έργο της σε σχέση με το μέλλον, να εξορίξει, να αντλήσει μαθήματα και συμπεράσματα από τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Eurojust στο παρελθόν και να τα προσαρμόσει για να μπορούν και στο μέλλον να αντιμετωπίζουν πιο εύκολα. Επιλογή βέλτιστων πρακτικών, best practices. Αυτά τα δύο είναι τα κύρια συμπεράσματα τα οποία εγώ συνάγω από τις πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Williams. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα όσον αφορά τα δύο αυτά ζητήματα. Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε. Ίσως η χρήση της αγγλικής δημιουργεί ε, κάποια σύγχυση, διότι από ό,τι καταλαβαίνω η λογοδοσία, το accountability, δεν μεταφράζεται ε, απόλυτα σε άλλες γλώσσες. Ίσως λοιπόν καλύτερο θα ήταν να μιλάμε για εποπτεία των δραστηριοτήτων και αυτό συμπεριλαμβάνει όλα όσα είπε ο συνάδελφος Εντία Τεμέρα. Θα πρέπει να γίνει η διάκριση ανάμεσα αυτού του τύπου την εποπτεία και τον έλεγχο, διότι ο έλεγχος ε, χρησιμοποιείται μόνο με την έννοια της εξέτασης συγκεκριμένων υποθέσεων και δεν είναι, αυτή η έννοια, δεν είναι αυτός, αυτού του είδους ο έλεγχος που θέλει να έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα πρέπει να εξετάσουμε μηχανισμούς ε, ώστε περιπτώσεις ε, όπου περιπτώσεις θυμάτων να μπορούν να εξεταστούν από ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από Εθνικά Κοινοβούλια. Όσον αφορά τον ε, Ευρωπαίο Εισαγγελέα, για να απαντήσω στον συνάδελφο Γιάν Μούλτερ, ε, νομίζω ότι τουλάχιστον στην τελευταία θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υπήρχε αρκετή υποστήριξη για την ιδέα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Μέχρι στιγμής όμως έχουμε ε, συναντήσει την, επιφύλαξη, την επιφυλακτικότητα των κρατών μελών όχι μόνο για αυτό το θέμα αλλά και για τις δραστηριότητες της Eurojust και της Europol και την, ε, το να τους δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες και για να μιλάμε για Ευρωπαίο Εισαγγελέα θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και δημοσιονομικό. Κοιτώντας το τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα, δεν καταφέραμε ούτε να λύσουμε το θέμα της ε, σύγκρουσης ε, δικαιοδοσιών λόγω των διαφορετικών ε, συμφερόντων των κρατών μελών. Και όταν κοιτάμε τις δραστηριότητες της Eurojust, να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Όταν μιλάμε για κοινέ ερευνητικέ ομάδες, εάν δείτε πώς υιοθετήθηκε η απόφαση όταν τροποποιήθηκε, αρχικά δώσαμε περισσότερες αρμοδιότητες στη Eurojust. Δώσαμε αρχικά περισσότερες αρμοδιότητες στην Eurojust με τη δημιουργία κοινών ερευνητικών ομάδων και τελικά καταλήξαμε στο να μπορεί να ελέγχει και να εγκρίνει κάθε φορά τη δημιουργία τους. Θέλω να πιστεύω ότι όταν δούμε πώς θα κινηθούν τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο όσον αφορά την, το, τη, την χορήγηση αρμοδιοτήτων ε, σχετικά με τη διεξαγωγή ερευνών. Πιστεύω ότι τότε θα είμαστε σε καλύτερη θέση να εκτιμήσουμε το αν το Συμβούλιο θα δεχτεί την ιδέα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Ευχαριστώ κύριε Τεφρέν. Πρόεδρε, τελικά βλέπουμε βαθμό το θέμα αυτό είναι κατεξοχήν πολιτικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα ευαίσθητο. Επιτρέψτε μου μια κάπως αφελή παρατηρήση. Μπορούμε να συζητούμε και να εμβαθύνουμε σε επίπεδο Υπουργών Δικαιοσύνη για τα θέματα αυτά. Όμω για το θέμα τη ποινική δικαιοσύνη στην Ευρώπη και το να εγκαταλείψουν τα κράτη ένα μέρο τη κυριαρχία του, βλέπουμε ότι το θέμα αυτό τελικά δεν έχει συζητηθεί επαρκώ διότι πραγματικά βλέπουμε πόσο αυτό συναρπάζει τους συνομιλητές και πόσο τεράστια προβλήματα θα υπάρχουν σχετικά. Ε, λυπάμαι που ακούω κάποιες παρεμβάσεις εδώ που μιλούν ε, για την αυστηρή εθνική κυριαρχία ε, και Ακούω να λέγεται ότι δεν πρέπει να υποκατασταθεί η εθνική εισαγγελία από την ευρωπαϊκή και ο καθένα θα πρέπει να μείνει στην ε, δική του την ε, μεριά. Τι πολιτική βούληση όμω τελικά έχουμε, τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον. Θέλουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο και το λέω αυτό ότι δεν μπορούμε να το σχεδιάζουμε κάτι τέτοιο χωρίς τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Εισαγγελικού σώματος. Το είπε όμως και ο Έλληνας συνάδελφος σωστά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα ποινικό δικαστήριο ε, με ανάλογες αρμοδιότητες. Ε, νομίζω λοιπόν ότι κάποιος έθεσε το θέμα των προδικαστικών ερωτημάτων και του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Βεβαίως ε, η συνθήκη της Λισαβόνας υφίσταται, λειτουργεί και ε, καταδεικνύει ότι ένα τέτοιο εισαγγελικό σώμα θα μπορούσε να σχεδιαστεί και να αρχίσει να γεννάται. Ε, εδώ λοιπόν ο ρόλος της Eurojust, το είπα και προηγουμένω ολοκληρώνοντα ότι θα βρει τη θέση που του αρμόζει. Αλλά το βασικό ζήτημα που θα μας αποσχολήσει τα ερχόμενα χρόνια, γιατί η πορεία αυτή θα είναι βραδία, είναι ένα θέμα πολύ ευρύτερο για το ποιο θα είναι το πραγματικό ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο, με όλα όσα προποθέτει. Διότι δεν μπορεί να υπάρχει δίκαιο χωρί κυρώσει βεβαίω, χωρί ποινέ. άρα οι κυρώσει, η εφαρμογή δηλαδή του δικαίου θα πρέπει να έχει πρεκοδοτηθεί και με μέσα προκειμένου να μπορεί να ασκηθεί σωστά. Ευχαριστούμε κυρία Ντεφρένια. Και τώρα νομίζω ότι έχουμε παραμένει στα πλαίσια του χρόνου. Σας ευχαριστώ όλους. Κλείσαμε με την τρίτη ομάδα ομιλητών και αμέσως περνάμε στην τέταρτη ομάδα ομιλητών. Προσκαλούμε τους ε, ομιλητές να έρθουν ε, στο Προεδρείο. Ο κύριος Γκούντερ Σόπενς από τη Βελγική Προεδρία ο κύριος Κοέλιου και η κυρία Σκοφιέ. Αγαπητοί βουλευτές, θα ξεκινήσουμε τώρα με την τέταρτη συζήτηση που έχει να κάνει με το πού ξεκίνησαν όλα. Μιλάμε εδώ για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Όλα αυτά, όλη η ιδέα αυτή ξεκίνησε του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ε, όλα αυτά λοιπόν ξεκίνησαν πριν 25 χρόνια με την, ε, με το, με την ιδέα του Σέγγεν. Έχουμε λοιπόν την 25η επέτειο της Συμφωνίας Σέγγεν που υιοθετήθηκε στην ομώνυμη πόλη στο Λουξεμβούργο τότε, αν δεν κάνω λάθος, ε, υπέγραψαν πέντε κράτη-μέλη. Από τότε ο χώρος Σέγγεν διευρύνεται συνεχώς και σήμερα περιλαμβάνει και χώρες εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, την Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ελβετία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Η ιδέα αυτή αναπτύσσεται συνεχώς από τότε. Και έχουμε εδώ του ομιλητέ μα που θα συζητήσουν το θέμα αυτό. Έχουμε τον κύριο Κούντερ ε, Κρέπεν που είναι πρόεδρος της ε, ομάδα Εργασία για, την αξιολόγηση, για τι αξιολογήσει Σέγγεν τη Βελγική Προεδρία. Θα πάρει πρώτο το λόγο. Κατόπιν θα πάρει το λόγο ο κύριος Κάρλος Κοέγιο, εισηγητής μας ε, σχετικά με το Σέγγεν στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατόπιν έχουμε την κυρία Αν Μαρή Εσκοφιέ που είναι γερουσιαστής στην Γαλλική Γερουσία. Κύριε Κόιπενς, έχετε το λόγο. Θα σας παρακαλούσα να περιοριστείτε σε ένα δεκάλεπτο. Θα το εκτιμήσω ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα. Είναι το ονομά μου. Είναι το όνομά μου Εργάζομαι για το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων στο Βέλγιο. Κατά τη διάρκεια τη ε, Βελγική Προεδρία, όπω αναφέρεται. Είμαι επικεφαλή τη ομάδα εργασία για την αξιολόγηση Σέγγεν. Κατά την παρουσίασή μου 10 λεπτών θα παρουσιάσω μια σύντομη εισαγωγή, θα σας δώσω μια επισκόπηση του χώρου Σέγγεν υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Συμβουλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μηχανισμό αξιολόγησης πέρα από τις δράσεις ε, Σέγγεν. Όπως προανέφερα το 1985, πέντε χώρες, ε, η Γαλλία, η Δυτική Γερμανία, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα αναμεταξύ τους. Σήμερα αυτός ο χώρος Σέγγεν αυξήθηκε σε ένα μεγάλο αριθμό κρατών μελών. Η ελευθερία κυκλοφορίας διασφαλίζεται για αυτά τα κράτη. Η Ελβετία, όπως επίσης αναφέρεται, είναι το πιο πρόσφατο μέλος του χώρου Σέγγεν προσχώρησε κατά τα τέλη 2008. Υπάρχει μια ιδιόμορφη κατάσταση για χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Δανία, με opt in και opt out εξαιρέσεις και συμμετοχές. Δεν θα επισέλθω περισσότερο σε αυτό το σημείο σήμερα. Πέρα από αυτά, ο χώρο Σέγγεν επίση συμπεριλαμβάνει κάποιε χώρε που δεν είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω η Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία. Ο τελικό στόχο για να δημιουργηθεί ένα χώρο χωρί εσωτερικά σύνορα είναι να επιτευχθεί και να είναι η πραγματικότητα ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται ένα υψηλό βαθμό ασφάλεια σε αυτό το χώρο. Πολύ πρόσφατα η σημασία μετακίνησης χωρίς φραγμούς τονίστηκε μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος στο Χόλμης και στις συνθήκες Λισαβόνας. Η Ένωση, αναφέρω παράθεμα, θα είναι ένας χώρος ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας με σεβασμό για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις διαφορετικές παραδόσεις ε, και έθιμα και συνήθειες των κρατών μελών. Έτσι έχουμε πάρα πολλά ωφέλη, όπως την υλοποίηση ενός ομοιογενούς χώρου ελευθερία και ασφάλεια χωρί εσωτερικά σύνορα. Όμω ε, ξεπερνά το πλαίσιο τη άρση των εσωτερικών σύνορων η δημιουργία μια κοινή βάση δεδομένων η διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία και η δικαστική συνεργασία καθώς επίσης ε, και η κοινή θεώρηση διαβατηρίων Σέγγεν για όλους όσους υπόκεινται σε αυτήν και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Θα ήθελα hm, αυτή τη στιγμή να επικεντρωθώ στα υπόλοιπα εννέα λεπτά που έχω στη διάθεσή μου μια, να σας δώσω μια επισκόπηση για το μηχανισμό αξιολόγησης ε, που ισχύει από το 1998 και πιο συγκεκριμένα τον ρόλο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ομάδα εργασίας αξιολόγησης Σέγγεν και το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα σχετικά. Αυτός ο μηχανισμός αξιολόγησης έχει δύο κυρίους στόχους αφενός να διοργανώνει αξιολογήσεις για κράτη υποψήφια προς ένταξη στο χώρο Σέγγεν, όπως για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, για παράδειγμα σήμερα. Αυτές είναι αξιολογήσεις υπό την πρώτη εντολή, first mandate. Και από την άλλη πλευρά να γίνονται αξιολογήσεις ώστε να διασφαλίζεται και να διαπιστώνεται αν τα μέλη του χώρου Σέγγεν εξακολουθούν να συμμορφώνονται και να υλοποιούν το και εκτιμένο του Σέγγεν. Και τέτοιου είδου ε, έλεγχοι ε, όσον αφορά τα ε, σύνορα, αν γίνονται με το σωστό τρόπο, αυτέ οι αξιολογήσει είναι αξιολογήσει δεύτερη εντολή, second mandate evaluations. Ο χώρο Σέγγεν βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη σίγουρα τα κράτη-μέλη έχουν άρει του ελέγχου στα εσωτερικά του σύνορα. Καταργούνται τα εσωτερικά σύνορα. Πρέπει όμω να υπάρχουν πιστικά οι έλεγχοι που είναι αποτελεσματικοί στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλίζονται τα άλλα κράτη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι στην ίδια αρχή τη αμοιβαία εμπιστοσύνη βασίζεται αυτό και έχουμε έτσι ομότιμα, ίσως ίσου προς ίσον τέτοιου τέτοιου peer to peer και είπα ότι υπάρχουν αυτές οι αξιολογήσεις από το 1998. Τότε η Εκτελεστική Επιτροπή είχε ε, θεσπίσει την μόνιμη επιτροπή όσον αφορά την αξιολόγηση της, ε, ε, των δραστηριοτήτων Σέγγεν και είχε και μια σαφή εντολή που μπορεί να βρεθεί σε αυτό το έγγραφο SCH κάθετος Connex 9826. Εκεί μπορείτε να βρείτε την σαφή εντολή για αυτού του είδους ε, της δράσης Schengen. Έχουμε επίσης και την ένταξη στο κοινοτικό κεκτημένο του κοινοτικού κεκτημένου, του κεκτημένου του Schengen και την μόνιμη επιτροπή που δημιουργήθηκε το προηγούμενο έτος που εντάχθηκε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι εντάχθηκε στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου. Εφ' εξής, ε, ο μηχανισμός ε, βρίσκεται υπό την αξιολόγηση της ε, Schengen Working Party, της ομάδας εργασίας αξιολόγησης Schengen, που είμαι πρόεδρος της. Και έχουμε επίση και την Coreper και το, στο Συμβούλιο που λογοδοτούν με εκθέσεις. Τι κάνουμε. Σε σχέση με τη δεύτερη εντολή έχουμε ένα μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων που προβλέπονται. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, το 2010 εφέτος έχουμε αξιολογήσει την Αυστρία, την Ιταλία και την Ελλάδα αξιολογήσει Ισπανία και Πορτογαλία βρίσκονται υπό εξέλιξη. Αυτέ είναι αξιολογήσει τη δεύτερη εντολή. Στην πρώτη εντολή, first mandate, έχουμε αξιολογήσει Ρουμανία και Βουλγαρία και αξιολογήσει του Λίχτενστάιν που θα διοργανωθούν πιθανότητα και θα λάβουν χώρα εφέτο. Επίση, όσον αφορά τι σκανδιναβικέ χώρε, Nordic countries, θα αξιολογηθούν Δανία, Φιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και είχαμε και πέσει την Γαλλία, Γερμανία και τι χώρε Μπενελούξ που αξιολογήσαμε. Έτσι λοιπόν μήνε πριν αρχίσουν οι αξιολογήσει, οι χώρε που βρίσκονται υπό αξιολόγηση πρέπει να απαντήσουν ένα εκτενέ ερωτηματολόγιο και να διαθέσουν όλα τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία. Αυτό είναι η βάση για τη δημιουργία ενό προγράμματο αξιολόγηση, για να ξεκινήσει η αξιολόγηση στη συνέχεια μετά. Υπάρχουν 7 κεφάλαια που εμπεριέχονται στι διαδικασίε αξιολόγηση. Αυτό σημαίνει γενικά ότι 7 προγράμματα αξιολόγηση συντάσσονται και πρέπει να γίνουν. 7 ομάδε αξιολόγηση αποστέλλονται και 7 εκθέσει αξιολόγηση συντάσσονται για κάθε χώρα. Είπα γενικά και αυτό φυσικά επειδή δεν έχει ε, νόημα να διοργανώνει κανείς ε, ε, αξιολογήσεις θαλασσίων συνόρων για μια χώρα που είναι μεσογειακή όπως η Αυστρία για παράδειγμα ή να γίνεται οτιδήποτε το αντίστροφο. Στα επτά κεφάλαια τα οποία αναφέρονται στις αξιολογήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, αξιολόγηση αστυνομικής συνεργασίας, αξιολόγηση χερσαίων συνόρων, θαλασσίων συνόρων, θέμα ε, χορήγησης διαβατηρίων, αξιολόγηση επ' και αξιολόγηση επίσης ε, της ε, αίτηση και συμμετοχής στο σύστημα πληροφοριών Schengen, Schengen Information System, SIS, SIS. Προεδρεύει έτσι λοιπόν η Συμβουλία και έχουμε και την γραμματεία της, ε, του Συμβουλίου, τη Γενική Γραμματεία. Υποβάλλονται τα στοιχεία αυτά και διατίθενται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το πρόγραμμα, πρόγραμμα αξιολογήσεων, πρέπει να προσαρμόζεται από το Schengen Evaluation Working Party, το, ε, την ομάδα εργασίας αξιολογήσεων του Schengen. Όταν έχει υιοθετηθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, αποστέλλεται εντολή προς τους επαείοντες των κρατών μελών που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτέ τι και τέτοιου είδους επαΐοντες σε σχέση με τις αξιολογήσεις διαφέρουν στη σύνθεσή τους από αξιολόγηση σε αξιολόγηση. Σε αξιολόγηση συνόρων υπάρχουν επαΐοντες μεταξύ 12 ή 15 για παράδειγμα. Ένα παράδειγμα αξιολόγηση του ΣΥΣ που έχουμε 5 ή 6 που συμμετέχουν. Το πρόγραμμα αξιολόγηση συντίθεται από διαφορετικέ ε, παρουσιάσει και εισαγωγέ. Όμω το πιο σημαντικό τμήμα τέτοιων αξιολογήσεων είναι οι επισκέψει επιτόπου όπου οι επαΐοντες μπορούν να αξιολογήσουν και να διαπιστώσουν πώς και σε ποιο βαθμό συμμορφώνεται κάθε χώρα εκάστοτε με το κεκτημένο του Σέγγεν. Η βάση αυτών των αξιολογήσεων αφενός ε, λαμβάνουν υπόψη το κεκτημένο Χάρτς, Συμφωνία του 1985, Σύμβαση του Σέγγεν, Σύμβαση ε, για θεωρήσεις διαβατηρίων Σέγγεν και το Soft Acquis. Το Hard Acquis και το ε, Soft Acquis, το σκληρό κεκτημένο και το ήπιο κεκτημένο. και και βιώματα από προηγούμενες δράσεις. Στο τέλος κάθε, μηχανι... Ε, κάθε ε, ε, αξιολόγησης μια έκθεση συντάσσεται, διαπιστώνονται ελλείψεις, διατυπώνονται συστάσεις, βέλτιστες πρακτικές αναφέρονται που μπορούν να είναι και υπόδειγμα για άλλα κράτη-μέλη. Έτσι οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται και σε κάποιες ελλείψεις όπως για παράδειγμα για τα όσα έχουν διακριβωθεί στα σύνορα. Υποβάλλονται αυτές οι εκθέσεις και συζητώνται από την ομάδα αξιολόγησης Schengen και με βάση αυτή την έκθεση η αξιολογούμενη χώρα συντάσσει ένα follow-up, μια συνέχεια σε έγγραφο όπου βελτιώσεις μπορούν να επιτευχθούν με βάση αυτές τις συστάσεις όσον αφορά οι λήψεις από την ένταξη 7 νέων κρατών από το 2007 έγιναν βελτιώσεις στο μηχανισμό αξιολόγησης και υπό την Γαλλική και Τσεχική Προεδρία για παράδειγμα έγιναν βελτιώσεις που αφορούν την προπαρασκευή του μηχανισμού αξιολόγησης και τον ίδιο τον μηχανισμό αξιολόγησης αφέ αυτού. Και υπό τη Βελγική Προεδρία τώρα κάποιες περαιτέρω βελτιώσεις γίνονται όσον αφορά τις διαδικασίες follow-up συνέχισης. Ολοκληρώνοντας θέλω να αναφέρω κάποια θέματα για το μέλλον προσβλέπουμε, στρέφουμε το βλέμμα προς το μέλλον και προσβλέπουμε τροποποιημένες προτάσεις Ευρω... Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα συμπληρώσουν τον υφιστάμενο μηχανισμό Σέγγεν που θα μπορούσαν να συζητηθούν από τον Νοέμβριο και εφ' Αναμένουμε λοιπόν αυτές τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στους επόμενους μήνες θα έχουμε ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, πράγμα το οποίο θα είναι σημαντική υπόθεση. Θα είναι μια ευκαιρία να συγχρονιστούν τα σύνορα της περιοχής Σέγγεν με τα, ε, τις ε, συνοδικές περιοχές αυτών των χωρών χωρών. Ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό είναι η δημοκρατική λογοδοσία στον χώρο ελευθερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Είμαι πεισμένο ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαζόμαστε μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, πράγμα το οποίο θα δίνει δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου αφενό, αλλά δεν θα δημιουργεί τριβέ και προσκόμματα και προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια αφετέρου. Με αυτόν τον τρόπο, ε, με αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να πω ότι μόνο όλοι από κοινού μπορούμε να συνεισφέρουμε για να επιτευχθεί αυτό ο στόχο για την Ευρώπη. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ. Τώρα, από πλευρά εισηγητού, από πλευρά ε, τη ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, θα έχουμε τον κύριο Κάρλο Κοέλιο που θα κάνει την παρουσίασή του, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρετίζω όλου του ε, συναδέλφου τη Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και του ε, βουλευτέ των Εθνικών Κοινοβουλίων και κυρίω ένα ιδιαίτερο χαιρετισμό στον κύριο Βουλευτή από την Πορτογαλία, τον κύριο Πεσότου, χώρα μου βεβαίω. Να πούμε λοιπόν ότι με 25 χρόνια του Σέγγεν θα θέλαμε να εξετάσουμε τη γέννησή του, το πώς εξελίχθηκε και τι επιτυχίε του. Ε, τώρα, οι επιτυχίε, λοιπόν ακριβώ αυτέ, τα 25 χρόνια. Πριν από 25 χρόνια, πέντε κράτη-μέλη αποφάσισαν να δημιουργήσουν, να προχωρήσουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ε, έροντα τα εσωτερικά του σύνορα και δημιουργώντα το χώρο Σέγγεν ανταποκρίθηκαν έτσι στα επικριτικά σχόλια τα οποία εξέφραζαν τη δυσαρέσκεια ότι τα κεφάλαια, τα αγαθά και οι υπηρεσίε είχαν μεγαλύτερη ελευθερία κυκλοφορία από ό,τι τα άτομα, οι πολίτε. Έτσι λοιπόν το Σέγγεν σημαδεύει την εξέλιξη τη ευρωπαϊκή αγορά, τη εσωτερική αγορά ε, προ την Ευρώπη των πολιτών, ε, την Ευρώπη των ανθρώπων. Η συμφωνία του Σέγγεν ήταν μια από τι μεγαλύτερε επιτυχίε τη ευρωπαϊκή ιστορία με την έμπνευση την ίδια των άλλων κοινών πολιτικών και την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Επίσης μας οδήγησε στην καλύτερη αντιμετώπιση των εγκλημα... της διασυνορικής ε, εγκληματικότητας με αστυνομή αστυνομικό και δικαστικό σώμα, οδηγώντας τη δημιουργία οργανισμών όπως η Eurojust και η Europol. Επίσης και η οικονομική στήριξη του χώρου Σέγγεν ε, υποβληθήθηκε από το Ταμείο ε, της ε, το Ταμείο του χώρου Σέγγεν και επίσης αφορά 400 εκατομμύρια πολίτες καθώς και 42.000 σύνορα χερσαία και θαλάσσια. Μάλιστα, σύντομα χώρο Σέγγεν μπορεί να αυξήσει, να τα μέλη του σε 28 με την συμμετοχή της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και του Λιχτενστάιν. Διευκόλυνε λοιπόν την κυκλοφορία των πολιτών, προώθησε την, τον τουρισμό και το εμπόριο και επέτρεψε του λαού της Ευρώπη να έρθουν πιο κοντά. Ωστόσο, αυτή και η ελευθερία της κυκλοφορία σημαίνει ότι υπάρχει και αύξηση των ευθυνών και τη ανάγκη κοινών αποκρίσεων παρόλο που κάθε κράτο μέλο έχει ακόμη την ευθύνη να ελέγχεται εξωτερικά του σύνορα ανάλογα με την επικράτειά του, ωστόσο αυτό το κάνει εξ ονόματο όλων των κρατών τη Ένωση, απαιτώντα να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν ε, πλήρως και αυστηρός ε, τα συνοδευτικά μέτρα ως προς την άρση των εσωτερικών συνόρων. Πράγματι, η ασφάλεια στον χώρο του Σέγγεν εξαρτάται από την αυστηρότητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία κάθε κράτος μέλος ελέγχει τα εξωτερικά του σύνορα. Επίσης και από την ποιότητα και την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, ο ευαίσθητο χαρακτήρα, η ανεπάρκεια στη λειτουργία, οποιοδήποτε από αυτού του παράγοντε ουσιαστικά θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ολόκληρη τη Ένωση και την αποτελεσματικότητα του χώρου Σέγγεν συνολικά. Παραλλήλω, η έκδοση ομοιόμορφων θεωρήσεων Σέγγεν από τα κράτη-μέλη επιτρέπει την στενότερη συνεργασία σε δικαστικό και αστυνομικό επίπεδο με τη στήριξη φορέων, εργαλείων και οργανισμών κοινοτικών προκειμένου να υπάρχει αυξημένο επίπεδο ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα, τα κοινά. Τώρα, για την κοινοτικοποίηση του Σέγγεν. Η διακυβερνητική συνεργασία προχώρησε. Όχι μόνο ε, λόγω αριθμού χωρών που συμμετέχουν, αλλά και από την θεσμική αρχιτεκτονική δομή. Ε, με την ε, συνθήκη του Άμστερνταμ το 1999 ε, εντάχθηκε στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το χώρο του Σέγγεν. Επίσης υιοθετήθηκαν κοινοτικά εργαλεία που αντικατέστησαν τους παλιούς κανόνες Σέγγεν όπως ο κώδικας συνόρων του Σέγγεν που ρυθμίζει τον έλεγχο των πολιτών στο πώς διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα, δίνει ένα κοινό πλαίσιο για τις αρχές και τους φορείς που ασχολούνται ακριβώς με τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν βελτιώσεις για όσους παίρνουν από τα σύνορα της Ένωσης, όμως περιορίζεται και η αρχική τάση απόλυτου ελέγχου που προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση Σέγγεν για την προσωρινή επανεισαγωγή των εσωτερικών σύνορων. Επίσης υπάρχει και ο κοινοτικός ε, κώδικας θεωρήσεων με βασικό στόχο να ελέγχεται η έκδοση των ε, ε, θεωρήσεων καθώς και οι αποφάσεις άρνησης, παράτασης, ακύρωσης, ανάκλησης, μείωσης διάρκειας της ε, διάρκεια των θεωρήσεων. Οι κοινέ προξενικέ οδηγίε ορίζουν ένα σύνολο κανόνων για τι θεωρήσει σύντομη διάρκεια με τη συνθήκη του Άμστερνταμ όπου, χαρακτηρίστηκε, όπου καθορίστηκε ο εμπιστευτικό του χαρακτήρα. και από το 2006 ήρθαν και κατάλληλε συμπληρώσει με τα βιομετρικά στοιχεία που θα ενσωματωθούν στο ΒΙΣ. Τώρα το σύστημα πληροφορήσεων για τι θεωρήσει, ε, το ΒΙΣ μετά τη Eurodac ε, και το ΣΥΣ είναι ένα σύστημα πληροφοριών ε, που αφορά το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Θα αποτελεί ένα σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών για τα 25 κράτη-μέλη που θα επιτρέπει στις αρμόδιε εθνικέ αρχέ να εισάγουν, επικαιροποιήσουν και να ε, συμβουλεύονται τα στοιχεία αυτά ηλεκτρονικώ. Θεωρείται μια από τι βασικέ πρωτοβουλίε στο πλαίσιο των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που σκοπό έχουν να προωθήσουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Το ΒΙΣ θα βελτιώσει τη διαχείριση, την πολιτική διαχείριση των θεωρήσεων, την προξενική συνεργασία και τις διαβουλεύσεις μεταξύ των κεντρικών προξενικών αρχών, προκειμένου να αναχαιτήσει ε, ε, απειλές στην εσωτερική ασφάλεια και προκειμένου να εμποδίσει και την ε, θύρα θεωρήσεων ε, δηλαδή να αναζητά κανεί το πιο εποφελέ καθεστώ θεωρήσεων που θα τον διευκολύνει. Επίση, θα διευκολύνει την καταπολέμηση τη παραχάραξη, παραποίηση ταξιδιωτικών εγγράφων, τον έλεγχο της μετανάστευσης και την παράνομη είσοδο στο, στην επικράτεια των 100 μελών, την επιστροφή των ε, λαθρομεταναστών. Με την εφαρμογή του κανονισμού Δουπλίνο 2 θα ε, ενισχυθεί η κοινοτική νομοθεσία σε σχέση με το άσυλο, οπότε θα αποτρέπονται και οι απειλές κατά της ε, κοινή εσωτερικής ασφάλειας και της τρομοκρατίας. Το σύστημα λοιπόν αυτή θα, αυτό θα επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο όσων περισσότερο στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Τώρα το σύστημα πληροφορίας του, ε, των θεωρήσεων, το ΒΙΣ τελικά μάλλον θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιούνιο του 2011 μετά από πολλέ καθυστερήσει. Τώρα το σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν από το 1999 είναι μεγαλύτερη και παλιότερη βάση δεδομένων στον τομέα τη εσωτερική ασφάλεια, των κοινωτικών. Ε, μιλάμε για διαδικτύωση των συστημάτων πληροφορική των ε, κρατών της, ε, του Σέγγεν όπου αποθηκεύονται τα στοιχεία αυτά από τις αστυνομικές και τελωνιακές αρχές των κρατών του Σέγγεν ε, με δυνατότητα συνεργασίας αστυνομικής και δικαστικής ε, ποινικά ζητήματα αλλά και τον έλεγχο των ανθρώπων που φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και θέλουν να περάσουν στην εθνική επικράτεια αλλά και την έκδοση θεωρήσεων. Η λειτουργία εδώ είναι διπλή. Η διατήρηση της ε, τάξης, της δημόσιας τάξης καθώς και η ασφάλεια σε επίπεδο μετανάστευσης να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών. Εδώ μιλάμε επίσης για έλεγχο ατόμων, ε, αντικειμένων και κλαπέντων οχημάτων. Οι σφαιρικέ κατηγορίε δεδομένων είναι όσοι αναζητούνται προ έκδοση, ε, επίση το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψη, οι πολίτε τρίτων χωρών ε, στου οποίου απορρίφθηκε η δυνατότητα εισόδου, οι αγνοουντες ε, άτομα και οχήματα τα οποία πρέπει να παρακολουθούνται ή συγκεκριμένες κατηγορίες ε, ε, απολεσθέντων ή εκλαπέντων αντικειμένων. Τώρα, το ΣΥΣ, η δεύτερη γενιά του ΣΥΣ, το ΣΥΣ 2, έχει και αυτό πέσει θύμα πολλών καθυστερήσεων. Ε, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα παρουσίασε πρόσφατα η Επιτροπή και θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα και οι λειτουργίε του ΣΥΣ2 θα ξεκινήσουν μόλι το 2013. Έπειτα το σύστημα ΣΥΣ θα συνεχίσει να λειτουργεί εντωμεταξύ με μια έκδοση που ονομάζεται ΣΥΣ One for All που βασικά είναι ένα κλόνο του εθνικού πορτογαλικού συστήματο και επιτρέπει στα κράτη-μέλη να συνδέονται στο κεντρικό σύστημα. Το ισχύον λοιπόν σύστημα ε, διέπεται από τους κανόνες της σύμβασης του Σέγγεν και το διαχειρίζεται η Γαλλία σε διακυβερνητική βάση. Το Ευρωκοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια ακολούθησε την κατεύθυνση της βασικής συμπερίληψης του συστήματος Σέγγεν στο ευρύτερο νομικό ευρωπαϊκό σύστημα, απορρίπτοντας οποιαδήποτε δυνατότητα να λειτουργεί ένα τέτοιο σύστημα σε διακυβερνητικό επίπεδο. Γι' αυτό στηρίξαμε τη δημιουργία του ΣΥΣ 2 και την δημιουργία νέου οργανισμού, προκειμένου να διαχειρίζεται όλα αυτά τα δεδομένα βάσει των νέων τεχνολογιών. Πέραν του τι σημαίνει το ΣΥΣ, ε, πέραν μάλλον από όλα τα υπόλοιπα. Το ΣΥΣ2 σημαίνει ε, μια αναβάθμιση τη ασφάλεια και τη ευελιξία μα στο σύστημα που χρησιμοποιούμε με την εισαγωγή βιομετρικών δεδομένων και την διασύνδεση των προειδοποιήσεων για τις απειλές. Αποτίμηση τώρα του Σέγγεν. Όπως είπε ο κ. Κέπενς που ε, προεδρεύει του ομάδα Σεβάλα όπως ονομάζεται, ομάδας αποτίμησης του Σέγγεν, υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα στην ουσία. Ένα σύστημα αποτίμησης ε, στην είσοδο και ένα σύστημα αποτίμησης για τα κράτη-μέλη που ήδη ε, συμμετέχουν στο σύστημα Σέγγεν. Η πρακτική μας εμπειρία μας έδειξε ότι είμαστε και τα περιορισμένοι στις φιλοδοξίες μας ε, και ε, επιτρέπουμε επίσης πολλά, είμαστε αρκετά επίοικείς ε, με όσα ανεχόμαστε. Ως προς τη χρήση του συστήματος Schengen, θα πρέπει να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναγγελία ότι φέτος θα δημοσιεύσει μια πρόταση σχετικά με τη δημιουργία ενός κοινοτικού μηχανισμού για την αποτίμηση του Schengen, πιο αποτελεσματικού, απλούστερου και πιο αποδοτικού, ώστε να υπάρχει διαφανής, ε, αποτελεσματική και συνεπής ε, υλοποίηση του χώρου Schengen. Επίση, το διακυβερνητικό πλαίσιο για την αποτίμηση του Σέγγεν θα προσαρμοστεί στο νέο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την ε, θέση σε ισχύ τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Γι' αυτό ακριβώ είναι καθοριστική σημασία να υπάρχει ένα συνεπή μηχανισμό αποτίμηση του Σέγγεν με συγκεκριμένε λειτουργίε οι οποίε αρχικά ε, ήταν διαιρεμένε μεταξύ πρώτου και τρίτου πυλώνα. Θα πρέπει όμω να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε εδώ για την ασφάλεια, για την ε, ασφάλεια στο χώρο δικαιοσύνη, ασφάλεια και ελευθερία. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών και από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπω ορίζουν οι συνθήκε, αλλά και από τα κράτη-μέλη, τα οποία συνεχίζουν βεβαίω να είναι αρμόδια για την ασφάλεια των εξωτερικών του συνόρων, εξού και η αρχή τη αμοιβαία εμπιστοσύνη, όπου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Τελευταίο θέμα, η διεύρυνση του Σέγγεν. Με την αποτίμηση των νέων κρατών μελών, όπω ήδη σχολιάστηκαν και σωστά τα ανέφερε ο κ. Κέπενς, με την δήλωση ικανότητας. Περιμένουμε ακόμη την αποτίμηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, αλλά μόλις όλα αυτά ολοκληρωθούν θα μπορέσουμε να δούμε αν θα υπάρξει και διεύρυνση του χώρου του Σέγγεν. Κλείνοντας, ε, Πρόεδρε, συνάδελφοι βουλευτέ, είναι ο σκληρό πυρήνα του χώρου ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη για μα, ο χώρο του Σέγγεν. Εδώ έχουμε το μεγαλύτερο επίπεδο ολοκλήρωση, αλλά χρειαζόμαστε και περισσότερα κοινωτικά εργαλεία, και παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, βλέπουμε ότι ο χώρο Σέγγεν είναι και καλύτερο, πιο αποτελεσματικό και υπάρχει και μεγαλύτερο συντονισμό. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστούμε κύριε Κοέλιο. Και τώρα η κυρία Ανμαρή Εσκοφιέ από την Γερουσία τη Γαλλία, παρακαλώ. Κυρίε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, 25 χρόνια μετά την υπογραφή στις 14 Ιουνίου του 1985 της Συμφωνίας του Σέγγεν, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το χώρο του Σέγγεν ως μια από τις μεγαλύτερες υποσχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είδαμε στα 25 αυτά χρόνια ε, ποιες ήταν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Οπότε από πέντε αρχικά κράτη-μέλη περάσαμε σχεδόν στο σύνολο των κρατομέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης δεχτήκαμε να δώσουμε και το καθεστώς σε χώρες, σε συνειδόμενα μέλη, σε τρία κράτη εκτός Ένωσης και που σύντομα θα γίνουν και τέσσερα. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η αρχική μας ε, σύλληψη για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών ουσιαστικά οδήγησε στην πραγματικά ελεύθερη κυκλοφορία και τους επακόλουθους στόχους. Έχουν, απαιτήθηκαν δέκα χρόνια βεβαίως για να υλοποιηθεί αυτή η κοινή βούληση και να καταργηθούν τα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των κρατών που επέγραψαν τη συμφωνία και να δημιουργηθεί βεβαίω και ένα οργανισμό για τα εξωτερικά σύνορα. Ελέγχεται έτσι η είσοδο στο χώρο Σέγγεν βάσει κοινών διαδικασιών που επιτρέπουν ελευθερία και δικαιοσύνη και την πρόθεσή του και βεβαίω διασφαλίζουν και το ευρωπαϊκό κοινό. Αυτά τα δέκα χρόνια βεβαίω, τα πρώτα δέκα χρόνια, ε, άλλαξε, ήταν μάλλον ένα διάστημα όπου άλλαξαν και η γεωπολιτική ισορροπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πτώση του τείχου του Βερολίνου, κατάρρευση του πρώην κομμουνιστικού καθεστώτο, πόλεμο των Βαλκανίων. Δέκα χρόνια όπου μετά την, ε, σύμβαση, την υπογραφή τη σύμβαση του Σέγγεν τέθηκαν σε ισχύ από το 1995 νέες μορφές τη συμφωνίας με εμβάθυνση το 1997 με το κεκτημένο του Σέγγεν και επίσης και το 2009 με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχουμε λοιπόν φτάσει 25 χρόνια μετά την πρώτη συμφωνία να είμαστε ισχυροί και να έχουμε ένα τεράστιο κληροδότημα στα χέρια μας. Ένα επίσης τεράστιο ε, τεκτημένο και νέους στόχους. Τώρα, να σταθώ στο εξής Πώς θα δημιουργήσουμε ένα κοινό σύστημα πληροφοριών, το σύστημα πληροφοριών Schengen, το SIS. Δεν ε, θα καθυστερήσω μιλώντα για το σύνολο μέτρων ε, που πολύ καλύτερα παρουσίασαν άλλοι πριν από μένα. Ήθελα απλώ να σταθώ στο πρόβλημα που δημιουργούν τα μέτρα αυτά σε δύο συγκεκριμένα σημεία. Πρώτα απ' όλα στην υλοποίηση των ε, αντισταθμιστικών μέτρων γενική εμβέλεια και επίση του δημοκρατικού ελέγχου, του ενισχυμένου δημοκρατικού ελέγχου του χώρου του Σέγγεν. Δύο λοιπόν προβλήματα τα οποία έχω ξεχωρίσει γιατί ακριβώς συζητήθηκαν επανειλημμένως στην Επιτροπή ε, του Κοινοβουλίου μας, όπου συμμετέ... της μάλλον, όπου συμμετέχω και εγώ. Τώρα, το σύστημα πληροφοριών ε, Σέγγεν. Είναι αυτονόητο ότι το να συντονίζει και να εναρμονίζει κανεί πολιτικέ δράσει ό,τι αφορά την εσωτερική ασφαλεία των κρατομελών δεν μπορεί να νοηθεί χωρί να υλοποιηθεί ένα σύστημα το οποίο το ίδιο να είναι συντονισμένο, εναρμονισμένο και να επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι πληροφορίε αυτέ είναι αναγκαίε και στι αστυνομικέ υπηρεσίε αλλά και στι δικαστικέ αρχέ, οι οποίε συμμετέχουν σε όλε τι διαδικασίε ελέγχου τη εισόδου και εξόδου από τα εσωτερικά εδάφη αλλά και τα εξωτερικά σύνορα τη Ένωση και για του πολίτες και για τα άγαθα. Το ΣΥΣ είναι ο καγωνιαίο λίθο, ε, ή μάλλον το θεμέλιο ε, αυτών των αντισταθμιστικών μέτρων. Είναι η βάση των δεδομένων λοιπόν που αποτελείται από, το κεντρικό, από τα κεντρικά συστήματα των κατομελών που έχουν διασυνδεθεί και επιτρέπουν να ανταλλάσσονται εθνικές πληροφορίες, ελεύθερη κυκλοφορία πληροφοριών, προκειμένου να λαμβάνονται τα επαραίτητα εθνικέ πληροφορίε, ελευθερη κυκλοφορια πληροφοριων προκειμενου να λαμβανονται τα επαραιτητα μετρα για την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών. Είναι ευαίσθητα δεδομένα αυτά τα οποία θα πρέπει να επακούν σε ένα διπλό στόχο. Αρκετά παράδοξο αυτό. Ότι θα πρέπει να δίνουν το μέγιστο δυνατό αριθμό πληροφοριών, προστατεύοντα όμω τον ιδιωτικό βίο των πολιτών. Για το θέμα αυτό έχω υποβάλει ήδη από πέρσι, με τη βοήθεια ενό συναδέλφου, μία πρόταση νομοσχεδίου, προκειμένου να προστατεύουμε καλύτερα τα προσωπικά δεδομένα και να προλαμβάνουμε, να, προλάβουμε μάλλον την αναθεώρηση τη ανάλογη Ευρωπαϊκή Οδηγία. Τώρα, η αύξηση του αριθμού των 100 μελών που χρησιμοποιούν το ΣΥΣ, καθώ και η τάση τη μεγαλύτερη χρήση τη πληροφορική οδήγησαν το 2001 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θελήσει να αναπτύξει ένα σύστημα δεύτερη γενιά, το ΣΥΣ 2. Ο κύριος Κοέλιο το ανέφερε προηγουμένως. Ένα σύστημα με νέες λειτουργίες, βελτιωμένο, το οποίο να βασίζεται στις νέες τεχνολογίες. Ωστόσο, το εγχείρημα αυτό ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί. Έχει καθυστερήσει λόγω τεχνικών αιτίων, που κυρίως έχουν να κάνουν με τον τεράστιο όγκο των νέων πληροφοριών που πρέπει να συλλεγούν. Ωστόσο, έχουμε δικαίωμα να αναρωτιόμαστε ποιε θα είναι οι συνθήκε χρηματοδότηση και οι τεχνικοί όροι που ε, οδήγησαν να θελήσουμε να περάσουμε από το ΣΥΣ στο Έχουμε μελετήσει αρκετά το σχέδιο προκαταρκτικά. Η διαχείρισή του είναι σωστή από την Επιτροπή που ανέλαβε την αρμοδιότητα αυτή με την εντολή του Συμβουλίου. Ε, η χρηματοδότηση είναι ρεαλιστική. Και αυτό εφόσον η Επιτροπή έχει εντοπίσει την ανάγκη να, να αποδοθούν 13 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην υλοποίηση του εγχειρήματο, που συνολικά θα κοστίσει 103 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν προβλέπονται στι ίδιε δαπάνε των κατομελών για τι εθνικέ του ε, επενδύσει. Βάσει του χρονοδιαγράμματο, το 2013 θα υπάρξει τέλο πάντων πλήρη μετανάστευση, όπω λέγεται, από το ΣΥΣ και το ΣΥΣ στο ΣΥΣ 2. Η Γαλλία από την πλευρά τη αμφισβητεί τι συνθήκε εντό των οποίων η πρώτη εξέταση και δοκιμασία, το τεστ του όλου συστήματο ξεκίνησε το 2010. Επιμένει η Γαλλία ότι το ΣΥΣ 2 θα πρέπει να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο επιδόσεων όπως και αξιοπιστία όπω το σημερινό σύστημα. Ω προ το Ευρωκοινοβούλιο ζήτησε έλεγχο από το ελεγκτικό συνέδριο για το σχέδιο αυτό ένας έλεγχος ορκωτός ο οποίο θα ολοκληρωθεί μόνο το 2011. Τώρα για τη δημιουργία οργανισμού διαχείρισης των συστημάτων πληροφοριών. Η διαπίστωση της Γαλλίας ε, ήταν ότι υπήρξαν δυσκολίε ε, με την υλοποίηση του ΣΥΣΔΙΟ Γι' αυτό η Γαλλική Γερουσία από το 2006 πρότεινε τη μεταφορά της διαχείριση του νέου συστήματο σε έναν αρμόδιο οργανισμό ad hoc του οποίου η έδρα να βρίσκεται στο Στρασβούργο. Στα πλαίσια όλου αυτού του προβληματισμού, η Σουηδική Προεδρία το φθινόπωρο του 2009 ξεκίνησε εργασίε για να δημιουργήσει ένα τέτοιο οργανισμό, ο οποίο ανέλαβε να διαχειρίζεται το σύνολο των συστημάτων πληροφοριών ε, μεγάλη εμβέλεια ό,τι αφορά το χώρο ελευθερία, δικαιοσύνη και ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή όλο ο προβληματισμό δεν μα έχει επιτρέψει να καταλήξουμε σε ένα χειροπιαστό σχέδιο που να ε, συμβάζει όλε τι προσδοκίε αλλά και τι δυσκολίε των κατομελών που συμμετέχουν. Ο καθένα, εφόσον έχει συνέστηση τη απόλυτη ανάγκη να υπάρχει ένα συνεπέ εργαλείο διαχείριση, ανάπτυξη ε, και διεύθυνση των ε, συστημάτων πληροφοριών, θα θέτει στον εαυτό του ερωτήματα για το ποιε είναι οι συνθήκε εντό των οποίων ε, θα αποτιμηθεί ένα τέτοιο σύστημα από το Συμβούλιο. Επίση, τίθενται ερωτήματα για τα δικαιώματα πρωτοβουλία τη Επιτροπή και των κρατών μελών, όπω θα διαμορφωθούν με τη δημιουργία ενό τέτοιου συστήματο. Ε, η απαραίτητη, ο απαραίτητος χρόνος για να περάσουμε σε ένα ΣΥΣ 2 αποτελεσματικό ε, προϋποθέτω ότι θα υπάρχει μια κοινώ αποδεκτή μεθοδολογία από όλου και προώθηση σωστών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ενισχυμένο δημοκρατικό έλεγχο. Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κοινοτική πολιτική. Η ανάπτυξη και η εκδίπλωση του χώρου Σέγγεν απαιτεί να υλοποιηθούν πολιτικές οι οποίες να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και την αυτοκυριαρχία των κρατών μελών. Είναι λοιπόν απολύτως αναγκαίο οι εκπρόσωποι των πολιτών, δηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια, να μπορούν να ασκήσουν έναν πραγματικό έλεγχο για τα μέτρα που υιοθετούνται. Η ανάγκη αυτή είναι μια διεκδίκηση της Γαλλικής Γερουσίας πολύ παλαιά. Επανειλημμένος το σώμα μας ε, τάχθηκε, υπέρ της δημιουργίας ε, ενός φόρουμ ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων με συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου για τον έλεγχο της Europol και της Eurojust. Να θυμίσω δύο εκθέσει συναδέλφων, του κ. Τούρκ και του κ. Τουρκουά που βρίσκονται εδώ μαζί μας, οι οποίοι ε, ζήτησαν τη δημιουργία ειδική επιτροπή όπου να συμμετέχουν ευρωβουλευτέ και εθνικοί βουλευτέ με την ευθύνη να παρακολουθούν τι δραστηριότητε τη Europol ακριβώ. Να πω ότι αυτή τη στιγμή στην Γαλλία ο συνταγματικό νόμο ε, του Ιουλίου 2008 παρέτεινε τι δυνατότητε έκφραση του Εθνικού Κοινοβουλίου επί των μέτρων που ε, υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικώς ποικιλία απόψεων μεταξύ ευρωβουλευτών και εθνικών βουλευτών δεν μπορεί παρά να αυξήσει το νόμιμον και το αξιόπιστο των, της παρακολούθησης των δράσεων από την πλευρά των πολιτών και για το πόσο υλοποιούνται τα μέτρα στο χώρο του Σέγγεν, που αφορούν το χώρο του Σέγγεν. Συμπερασματικό λοιπόν μπορούμε να εκφράσουμε ικανοποίηση για το πόσο αποφελήθηκαν από τις ε, συμβάσεις του 90 τα κατημέλη. Ο απολογισμός βεβαίως δεν είναι μόνον ικανοποιητικός, διότι τα 25 αυτά χρόνια επέτρεψαν στα κράτη μας που πλέον ζουν σε συνθήκες ειρήνης να ε, βρουν τρόπους ε, για να αντιμετωπίσουν κοινωνικά προβλήματα σε συνθήκε ασφάλειας. Προβλήματα όμως τα οποία θα βρουν την απάντησή τους σε μια ρεαλιστική και χειροπιαστή συνεργασία. Να μην ξεχνάμε ότι και η Ρουμανία με τη Βουλγαρία μπορεί να έρθουν μαζί μας από τον Μάρτιο του 2011 στο ίδιο πνεύμα συνεργασίας, με τις ίδιε αξίε, σε ένα κοινό χώρο ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη για όλους τους λαούς μας. Now we open Ευχαριστούμε. Ξεκινάμε τώρα τη συζήτηση. Ο κύριος Τσίποφ από το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, Τον Μάρτιο του 2011 ελπίζουμε ότι θα προσχωρήσουμε στον χώρο του Σέγγεν. Αυτό για μας αποτελεί προτεραιότητα. Έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα κλίμα άριστης συνεργασίας με, τους διάφορους, ε, με τα διάφορα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς που θα μας οδηγήσουν σε αυτό το στόχο και θέλουμε να υλοποιήσουμε όλους τους κανόνες Σέγγεν προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ασφαλή από το 2007 ως το 2010 έχουμε αναλάβει όλα τα τις απαραίτητες δράσεις προκειμένου να εναρμονίσουμε την δική μας εθνική νομοθεσία με το κοινοτικό κεκτημένο. να, να χρησιμοποιήσουμε τα απαραίτητα μέσα και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Έχουμε απευθύνει κλήσει στις υπόλοιπε χώρες, έχουμε υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές τους. Και χάρη στην πρωτοβουλία της βουλγαρικής κυβέρνησης, έχουμε παρατείνει τις ε, προθεσμίες και τις διάρκειες διαπραγμάτευσης προκειμένου να είμαστε στις καλύτερες δυνατές επιδόσεις τη στιγμή που θα προσχωρήσουμε και να μπορούμε να διαχειριστούμε και οποιαδήποτε κρίση. Ωστόσο, να πιστήσω την προσοχή σας στο εξή. Πολλές συμβάσεις για τους εξοπλισμούς έχουν συναυθεί με άλλα κράτη-μέλη με συνολική αξία εκατομμύρια ευρώ από το 2008 στο 2010 και με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσαμε σε μία αυτοαξιολόγηση όπου διαπιστώσαμε κενά και ελλείψεις και φροντίσαμε να συμπληρώσουμε τα κενά και τις ελλείψεις αυτά με τα απαραίτητα μέτρα, να τις ξεπεράσουμε. Οι διάφορες σχετικές εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν από τους αρμόδιους εμπειρογνώμονες μας ενεθάρρυναν να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση για να επιτελέσουμε πρόοδο. Οι εκθέσεις αυτές βεβαίως περιλαμβάνουν και συστάσεις, συστάσεις βελτίωσης κάποιων πτυχών της δράσης μας. Καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών λόγου χάρη, καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων. Στις 29 Ιουνίου 2010 λοιπόν Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τους τελευταίους εφαρμοστικούς κανόνες του ΣΥΣ 2 ορίζοντας ε, τις διορίες ε, ενσωμάτωσης και συμπερίληψης του συστήματος αυτού και στο βουλγαρικό μεταξύ των υπολείπων. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι έχουμε προβλέψει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Έχοντας υπόψη και σεβόμενοι και τα ατομικά δικαιώματα και τους κανόνες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. Ελπίζουμε έτσι ότι θα μπορέσουμε να προσχωρήσουμε στο χώρο του Σέγγεν ήδη το Μάρτιο του 2020. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ένα πρωταρχικό ερώτημα. Η κατάργηση των συνόρων στα πλαίσια του ενιαίου χώρου Σέγγεν δημιουργεί πράγματι νέα δεδομένα και επί 25 χρόνια τώρα θεωρώ ότι πλανάται ένα θεμελιώδες ερώτημα. Η απελευθέρωση του χώρου που προκύπτει από την κατάργηση των συνόρων από ποιον καταλαμβάνεται από την κοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών ή από ένα θεσμικό ή υπερθεσμικό πλάσμα που θα μπορούσαμε και έχει αυτό ήδη πολλές φορές λεχθεί θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε ένα σύγχρονο Big Brother. Και θεωρώ επίσης μια βασική έλλειψη το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν διατυπωθεί όσο θα έπρεπε τα παράπονα εκείνα από τα κράτη-μέλη που έχουν να κάνουν με την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν μέχρι στιγμής και ακούγοντας τους προλαλήσαντες διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει κοινή συμφωνία, κοινή άποψη για το ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό σύστημα εκτίμησης των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία επί 25 χρόνια της συνθήκης του Σέγγεν. Αυτό ήδη θεωρώ ότι είναι μια αρνητική αξιολόγηση. Και θα πρέπει επιτέλους να πούμε και ένα τελικό λόγο επάνω σε αυτό μέχρι σήμερα. Σε τι μπορούμε να πούμε για τα κράτη-μέλη ή για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποδοθεί η έκφραση ότι αποτελεί η συνθήκη Σέγγεν και επί 25 χρόνια λειτουργία της τον ακρογωνιαίο λίθο ή το σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα τουλάχιστον όσον αφορά τις προτεραιότητες επάνω στις οποίες θα πρέπει να στηριχθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά αν θέλετε και υπέρ της κοινωνίας των Ευρωπαίων πολιτών αναφορικά με τα πολύ συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τις διαδικασίες αυτές και αφορούν κυρίως την προστασία των πολιτών από φαινόμενα όπως είναι η διακίνηση των ναρκωτικών, όπως είναι η διακίνηση του μαύρου χρήματος, όπως είναι η διακίνηση ή η δράση οργανωμένων εγκληματικών οργανώσεων και βεβαίως οπωσδήποτε και της τρομοκρατίας. Σε αυτούς τους τομείς τι έχει αποδώσει η συγκεκριμένη λειτουργία του χώρου της Έγκεν και βέβαια θα έχω μια περιέργεια να μάθω η Ελβετία όσον αφορά τα προηγούμενα που ανέφερα κατά ποιο τρόπο μπορεί να θεωρηθεί ότι συμμετέχει ή λειτουργεί στα πλαίσια αυτού του ενιαίου χώρου όταν αρνείται συστηματικά να δώσει στοιχεία τα οποία αφορούν καταθέσεις ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με εγκληματικές πράξεις που προφανώς είναι εναντίον μιας δίκαιης και ασφαλούς και σε συνθήκες ελευθερίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. κύριε κύριος από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών της Ευρωβουλής. Σας ευχαριστώ. Și eu, la rândul meu, consider că Schengen este unul dintre cele mai puternice simboluri ale capacității. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσωπικά πιστεύω ότι η περιοχή Σένιεν είναι ένα από τα ε, σημαντικότερα σύμβολα της ικανότητας της Ευρώπης να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών μας. Όπως είπε και ο συνάδελφός μας κύριος Κοέλιο, είναι ένα ε, επιτυχημένο εγχείρημα που αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της Ευρώπης τα τελευταία 30 χρόνια. Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρώπης μπορεί να υπάρξει μόνο εάν υπάρχει ελεύθερη κινητικότητα των πολιτών. Το σύστημα αξιολόγησης Schengen είναι απλό, αποτελεσματικό και διαφανές. Σήμερα λοιπόν και στο μέλλον θα μπορούμε να ε, διασφαλίσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών καθώς και την ασφάλεια. Θα ήθελα να ε, ρωτήσω ε, την κυρία Εσκοφιέ το εξής. Πιστεύετε εσείς ότι τα πρόσφατα γεγονότα στη Γαλλία μπορούν να οδηγήσουν σε αμφισβήτηση του χώρου Σέγγεν. η γαλλική κυβέρνηση έχει προειδοποιήσει την ε, Ρουμανία ότι πιθανότατα δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην περιοχή Σέγγεν από, το, από την Άνοιξη. Μήπως αυτό έγινε βιαστικά, μήπως θα έπρεπε να έχει συζητηθεί το πράγμα στο Συμβούλιο πριν από τις δηλώσεις Τη Γαλλία. πριν προχωρήσει σε δηλώσει η Γαλλία και θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο ή ε, θα εξεταστεί απλά η έκθεση σχετικά με τη Ρουμανία. Ευχαριστώ κύριε Σέπτσικ από την γερουσία της Τσεχίας. Ευχαριστώ για τις αρχικές ομιλίες που ακούσαμε. Η Τσεχία είναι μία από τις τελευταίες χώρες που προσχώρησαν στον χώρο Σέγγεν. Πιστεύω ότι οι πολίτες μας είναι ικανοποιημένοι με αυτό. Υπάρχει εδώ ένα σημαντικό ψυχολογικό αποτέλεσμα. Όταν ταξιδεύει κανείς εκτός της χώρας του και δεν ελέγχεται στα σύνορα, νιώθει ότι ανήκει σε μια περιοχή. Οι Τσέχοι πολίτες βλέπουν ε, την ε, αυξημένη παρουσία τσέχων στις γειτονικές μας χώρες ε, λόγω της περιοχής Σένιεν. Θα πρέπει οι γειτονικές μας χώρες να αρχίσουν να μας εμπιστεύονται, να μην θεωρούν τους πολίτες μας επικίνδυνους για τις χώρες τους. Ωστόσο, κάποιες, κάποιοι έλεγχοι που γίνονται δεν σέβονται την αξιοπρέπεια των πολιτών μας. Εγώ ο ίδιος ε, ζήσα μια, ένα τέτοιο συνοριακό έλεγχο. Ένα αυτοκίνητο με σταμάτησε, με, πήγανε, με οδήγησαν σε ε, ε, ένα κτίριο κοντά στον αυτοκινητόδρομο και μου ζήτησαν να ανοίξω τις αποσκευές μου. δεν ήταν ευχάριστη η εμπειρία αυτή, ήταν ταξίδι για ιδιωτικούς σκοπούς. Δεν νομίζω ότι σέβονται την αξιοπρέπεια των Τσέχων πολιτών τέτοιοι έλεγχοι θα χαιρόμουν εάν δεν γίνονταν τόσοι τέτοιοι έλεγχοι. Καταλαβαίνω ότι είναι απαραίτητο να γίνονται κάποιοι τέτοιοι έλεγχοι. Ο τρόπο όμω με τον οποίο διεξάγονται δεν είναι σωστό. Ευχαριστώ κύριο Καϊσεύσκη. Από τη γερουσία τη Πολωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώντας, θέλω να πω ότι δεν μπορώ να κατανοήσω απόλυτα τα όσα είπε ο Έλληνα συνάδελφο. Τι είναι αυτό το οποίο επιθυμεί. Θέλει να αποκατασταθούν τα εσωτερικά ε, σύνορα των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εχθές κάναμε λόγο για την υπηρεσία Frontex που πιστεύω ότι όλο και περισσότερο αυξάνει ή ενδυναμώνει τον χώρο Σέγγεν και προστατεύει τα κοινά εξωτερικά μας σύνορα. Τώρα, η Πολωνία ενδιαφέρεται φυσικά από πλευράς της ώστε να διασφαλιστεί ότι θα έχουμε διασυνοριακή δυνατότητα κυκλοφορίας χωρίς θεωρήσεις διαβατηρίων μεταξύ Ολλανδίας μέχρι την ε, Λευκορωσία, ακόμα και μέχρι την, το Καλίνιγκρα, την αυτόνομη ρωσική περιοχή που συνορεύει ε, Τώρα αυτή η προσέγγιση νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντική υπό το πρίσμα της ελεύθερης κυκλοφορίας, υπό το πρίσμα της επικοινωνίας αναμεταξύ μας, διότι αυτό καθιστά τον χώρο Σέγγεν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την φέρνει πιο κοντά στις χώρες εκείνες που δεν μπορούν ακόμα σε αυτή τη φάση να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γειτονικέ μας χώρες. Έτσι ο χώρος Σέγγεν το καθιστά εφικτό για μας και είναι, το κάνει δυνατό να είμαστε πιο κοντά, να προσεγγίζουμε αυτές τις χώρες από πλευρά μα εμεί. Και πρέπει να είμαστε σε θέση να καταδείξουμε στου γείτονέ μα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το μέλλον του θα έπρεπε να είναι στην Ευρώπη και όχι στην Ασία. Ευχαριστώ. Και η κυρία Γιώτοβα στη συνέχεια της Επιτροπής Λίμπε. Euh, Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μία ερώτηση θα είχα που θα ήθελα να διατυπώσω Κύριε Καϊπενς, θα μπορούσατε ίσως να μας πείτε δύο λόγια για την Βουλγαρία και τη Ρουμανία διότι η ομάδα σας, η επιτροπή σας, ας το πω έτσι, ασχολείται ακριβώς με αυτά τα θέματα. Πώς έχει το πράγμα με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται. Καθυστερήσεις όσον αφορά την αξιολόγηση των κριτηρίων. Τι γίνεται σε σχέση με την ένταξη αυτών των δύο χωρών στο Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ένστα από την Επιτροπή Λίμπε, παρακαλώ. ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ουσιαστικά δύο πράγματα θα ήθελα να πω. Το πρώτο, επενέθηκε πολύ το Σέγγεν. Φυσικά το Σέγγεν δεν είναι τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω από ένα πλαίσιο, ας το πω έτσι, για τις χώρες ένα πλαίσιο για την ελευθερία της κυκλοφορίας και της διακίνησης. Πρέπει ρεαλιστικά να το δούμε αυτό. Πώς διαμορφώνουμε αυτό το πλαίσιο είναι το δεύτερο θέμα, το δεύτερο ερώτημα. Και όσον αφορά τις, τους ανθρώπους, αυτοί θέτουν το θέμα για τις συνθήκες διαβίωσής τους. Πώς βελτιώνονται, τι συνεισφέρει προς αυτό. Και ούτως ή άλλως, ναι μεν έχουμε με το Schengen ένα πλαίσιο, αλλά δεν έχουμε τη διαμόρφωση αυτού του πλαισίου τελεσίδικα. Αυτό θα ήθελα να πω. Και για να επανέλθουμε σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο ως ε, θέμα όταν τοποθετούμαστε σε τέτοια θέματα. Δεύτερο σημείο, SS2. Ξέρετε ότι είναι επίμαχο και για χρηματοοικονομικούς αλλά και για πολιτικούς λόγους πρέπει να προσθέσουμε αν δει κανεί ποια, ποια στοιχεία, ποια προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται και δεδομένα που αφορούν τις μυστικές υπηρεσίες κτλ. Ε, το εξή θα ήθελα να θέσω. Την προηγούμενη εβδομάδα η Επιτροπή Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε τα κονδύλια για την περαιτέρω εξέλιξη του SS2 να τα παγώσει. Δηλαδή τα κονδύλια για την εξέλιξη, μετεξέλιξη αυτού του SS2 δεν θα υπάρξουν αυτά τα κονδύλια. Υπάρχουν αμφιβολίες αν υπάρχει ένα ρεαλιστικό χρονοπλαίσιο στα χέρια μα στη διάθεσή μα. και μήπω έτσι διακυβεύονται κάποιε εξέλιξει. Ερώτησή μου, τι γίνεται σε σχέση με τις κυρίες και κυρίους στο Προεδρείο. Πώς βλέπετε εσείς τις περαιτέρω εξέλιξη του SES2 υπό, αυτές, υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτική για, αυτό το, για αυτή την εξέλιξη. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Ντάνοκα από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Πολιτικών Ελευθεριών. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε δρατώμενη της ευκαιρίας και εγώ θα ήθελα να διατυπώσω μία ερώτηση προς τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου και αφορά μια άλλη ίσως προσέγγιση προς το Σέγγεν, προς τον χώρο Σέγγεν σε σχέση με δύο κράτη υποένταξη που δεν είναι ακόμα ε, κράτη-μέλη, δηλαδή την Βρετανία και την Ιρλανδία. Δεν είναι κράτη-μέλη του Σέγγεν, ενώ είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε ούτε καν να εναρμονίσουμε απαιτήσει ε, για την διάβαση των συνόρων σε σχέση με την κατάσταση όπως υφίσταται σε αυτά τα δύο κράτη-μέλη και για τις θεωρήσεις διαβατηρίων. Όμως υπάρχουν κάποια βήματα που γίνονται από πλευρά του Συμβουλίου σε σχέση με αυτά τα δύο κράτη-μέλη για έναν εναρμονισμό αυτού του χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας ατόμων. Πρώτα απ' όλα το πρόβλημα τίθεται για τους μόνιμα διαμένοντες με μόνιμη άδεια εγκατάστασης για αυτά τα άτομα που έχουν την έδρα τους στην, στο χώρο Σέγγεν ενώ είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Υπάρχουν κάποια βήματα τα οποία γίνονται για να βελτιωθεί η κατάστασή τους όταν έρχεται η ώρα ελεύθερης κυκλοφορίας για αυτά τα δύο κράτη-μέλη, δηλαδή τη Βρετανία και την Ιρλανδία, για αυτή την κατηγορία ατόμων που έχουν άδεια εγκατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστροφα να περνούν στον χώρο Σέγγεν μόνιμοι κάτοικοι της Βρετανίας και της Ιρλανδίας. Ευχαριστώ. Και τώρα από πλευρά των όσων συμμετέχουν εδώ στο Προεδρείο θα πρότεινα με την ίδια σειρά όπως παρενέβησαν στον πρώτο γύρο. Ο κύριος Κόιπες πρώτος, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εάν υπάρχει Ολλανδικ... Ε, η μετάφραση θα μιλήσω Ολλανδικά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις παρατηρήσεις σας Πολλές τις ε, κατέγραψα και θα επανέλθω σε αυτές. Θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι που είπε ο κύριος Κοέλιο. Μίλησε για τις αξιολογήσεις των χωρών που θα γίνουν μέλη του Σένιεν. Η πρώτη εντολή, οι αξιολογήσεις πρώτης εντολής έχουν διεξαχθεί πολύ σοβαρά και το ίδιο ισχύει για τις αξιολογήσεις της δεύτερης εντολής. Για παράδειγμα, έγινε αξιολόγηση του Βελγίου και μπορώ να σας πω ότι έγινε πολύ σοβαρή δουλειά. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην παρατήρηση του Έλληνα συναδέρφου σχετικά με τα δεδομένα που χρειάζονται για τη συνεργασία στον ποινικό τομέα. Η ομάδα εργασίας μου έχει πολύ σαφή εντολή. Και στην εντολή της ομάδας μου δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποινικά θέματα. Δεν μπορώ λοιπόν να απαντήσω. Θα ήθελα να απαντήσω και σε μια ερώτηση που σημείωσα που έχει να κάνει με την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας και τις σχετικές προθεσμίες. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται εδώ και λίγο καιρό. Το τελευταίο κεφάλαιο που θα ε, πρέπει να αξιολογηθεί είναι το SIS, το Σύστημα Πληροφόρησης Σέγγεν. 6 με 12 Σεπτεμβρίου γίνεται η αξιολόγηση ε, για το κεφάλαιο αυτό και έτσι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία προσχώρησης. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια ερώτηση που αφορά την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν συμμετέχουν στο Σέγγεν. Υπάρχει μια σειρά θεμάτων που είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αποτελούν αποκλειστικά αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η εντολή της ομάδας εργασίας μας δεν μας επιτρέπει να πάρουμε θέση σε τέτοια ζητήματα. Δεν μπορώ λοιπόν να απαντήσω. Δεν μπορώ να απαντήσω δηλαδή σε ερωτήσει που έχουν να κάνουν με την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι δεν καλύπτονται από την εντολή μα. Ελπίζω να απάντησα στι ε, ερωτήσει, τουλάχιστον στι πιο βασικέ. Ο κύριο Κοέλιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρει παρατηρήσει. Ε, πρώτον, ε, να απαντήσω στον Έλληνα φίλο. Δεν Πιστεύω ότι ήταν κακή η απόφαση να έρθουν τα εσωτερικά σύνορα. Πιστεύω ότι ήταν καλό αυτό για την Ευρώπη, καλό για τους πολίτες, καλό για την ελευθερία, καλό για τον τουρισμό. Και πιστεύω ότι η ζωή θα ήταν πιο δύσκολη για τους Ευρωπαίους πολίτες εάν ε, ε, ξαναδημιουργήσουμε τα εσωτερικά σύνορα. Δεν νομίζω ότι αυτό θα ήταν σωστή απόφαση. Ούτε θα πρότεινα να συγκρίνουμε το σύστημα πληροφόρησης Schengen με τον μεγάλο αδερφό. Εάν κάποιος προσπαθήσει να εισέλθει στην ε, Πορτογαλία μέσα από εξωτερικά σύνορα, σημαίνει ότι εισέρχεται στη Γαλλία, στην Ισπανία, δεν υπάρχουν εσωτερικά σύνορα. Στα... Η αστυνομία στα πορτογαλικά σύνορα, λοιπόν, θα πρέπει να έχει πληροφορίες ε, για το πρόσωπο αυτό και να τι στείλει στα άλλα κράτη-μέλη, διότι τελείως δεν μπορούμε να διατηρήσουμε υψηλό επίπεδο ασφάλειας όπως επιθυμούμε. Πάντα βέβαια, όταν μιλάμε για σύγχρονη τεχνολογία και μεγάλες βάσεις δεδομένων, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ε, να δημιουργηθεί ένας νέος μεγάλος αδερφός. Γι' αυτό έχουμε αυστηρούς κανόνες όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους κανόνες που έχουμε υιοθετήσει και τον τρόπο που τους εφαρμόζουμε. Όσον αφορά τη δεύτερη γενιά του συστήματος πληροφόρησης Schengen, θα ήθελα να τονίσω, όπως ήδη υπόθηκε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει τη συγκεκριμένη γραμμή του προϋπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον θα ξεμπλοκάρουμε τη γραμμή ε, αυτή του προϋπολογισμού εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δώσει όλες τις πληροφορίες που ζητάμε. Κατά τη γνώμη μου χρειαζόμαστε τη δεύτερη γενιά του συστήματος πληροφόρησης Schengen. Το SIS-2 χρειάζεται για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για λόγους ασφαλείας. Σύντομα αναφέρθηκα στη συζήτησή μου, στην ομιλία μου σε αυτό. Πρώτον, ε, έχουμε βιομετρικά δεδομένα. Τώρα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στα σύνορά μα το λεγόμενο πρόβλημα John Smith. Όταν συλλαμβάνουμε κάποιον ή τον σταματάμε με... που έχει το ίδιο όνομα με κάποιον που ήδη βρίσκεται στο σύστημα, Εάν υπάρχει κάποιος Κάρλος Κοέγιο με κάποια καταχώρηση, με ε, ε, ένα σήμα συναγερμού στο σύστημα, ε, το σύστημα θα πει ότι «Α, είναι επικίνδυνος». Δεν είμαι όμως εγώ, είναι άλλος Κάρλος Κοέγιο. Εάν λοιπόν το ΣΥΣ έχει βιομετρικά δεδομένα, μπορώ με τα δακτυλικά μου αποτυπώματα να αποδείξω ότι δεν είμαι εγώ αυτός στο σύστημα για τον οποίο έχει γίνει ε, ε, αυτή η θετική καταχώρηση. Τα βιομετρικά δεδομένα λοιπόν είναι τρόπος να καταπολεμήσουμε ε, τις ψευδείς ταυτότητες και άλλα προβλήματα του συστήματος άλλος τρόπος να βελτιώσουμε την ασφάλεια είναι η διασύνδεση ανάμεσα στις θετικές καταχωρήσεις. Αυτή τη στιγμή, εάν υπάρχει κλεμμένο αυτοκίνητο, το μόνο πράγμα που μπορούμε να ρωτήσουμε το σύστημα είναι το αυτοκίνητο αυτό είναι κλεμμένο ή όχι. Δεν δίνονται όμως άλλες πληροφορίες. Εάν συνδέσουμε τις θετικές καταχωρήσεις, μπορούμε να συνδέσουμε το όχημα με κάποιο αυτοκίνητο ή με κάποια εγκληματική πράξη. Δεν είμαι αστυνόμικος, αλλά καταλαβαίνω ότι η με καποια εγκληματικη πραξη δεν ειμαι αστυνομικο αλλα καταλαβαινω οτι η προσεγγιση τη αστυνομία είναι διαφορετική. Ε, ανάλογα με το αν το όχημα αυτό είναι ένα απλό αυτοκίνητο ή ένα απλό κλεμμένο αυτοκίνητο ή αν συνδέεται με ένα δίκτυο ε, παιδοφιλίας ή τρομοκρατίας. Η προσέγγιση λοιπόν τη αστυνομία είναι διαφορετική στι δύο αυτέ περιπτώσεις. Τέτοιου είδου πληροφορίε θα παρέχονται από τη δεύτερη γενιά του συστήματο ΣΥΣ και γι' αυτό χρειαζόμαστε το ΣΥΣ 2. Και τελευταία απάντηση για τον συνάδελφο από την ε, Βουλγαρία. Βεβαίως, η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ε, στο χώρο Σέγγεν μας απασχολούν ιδιαίτερως. Εδώ στο Κοινοβούλιο είχα τη χαρά να υποδεχθώ τον ε, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης που είναι και υπουργός εσωτερικών της Βουλγαρίας και για το Ευρωκοινοβούλιο αποτελεί πολιτική προτεραιότητα το ζήτημα αυτό. Θέλουμε η Βουλγαρία και η Ρουμανία να συμμετέχουν στο χώρο του Σέγγεν, διότι ανήκουμε στην ίδια ευρωπαϊκή οικογένεια. Είναι δική μας πολιτική βούληση αυτή. Όμως, όταν μιλά κανείς για Σέγγεν, δεν αρκεί απλώς η βούληση, η πολιτική. Πρέπει να υπάρχει και το σεβασμό του συστήματος αποτίμησης. Και βεβαίω και για τη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου σε όλο αυτόν τον ε, μηχανισμό αξιολόγηση υπό την προεδρία του κυρίου Κιόπεν, που είδε και ένα μηχανισμό διακυβερνητικό. Τα κράτη-μέλη πρέπει να επαληθεύουν κατά πόσον οι συνθήκε υπάρχουν, ε, κατά πόσο πληρούνται όλα τα κριτήρια. Και αυτό πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα. Άρα, κυρίως για την Βουλγαρία και την Ρουμανία έγκυται η ευθύνη, το βάρος της ευθύνης, να αποδείξουν ότι είναι σε θέση, ότι είναι σε θέση να συμμετέχουν πλήρω στο χώρο Σέγγεν. Θέλουμε λοιπόν να έρθετε στην οικογένειά μα, αλλά πρέπει να βρίσκεστε στο δικό μα επίπεδο ασφάλεια. Διότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι απολύτω αναγκαία. Πρέπει να υπάρχει ε, βεβαιότητα ότι το είδο ελέγχων που διενεργούν η Βουλγαρία και η Ρουμανία στα ρουμανικά και βουλγαρικά σύνορα είναι ακριβώς της ίδια ποιότητα με όλων των κρατών μελών στα δικά του σύνορα. Ελπίζω λοιπόν ότι η αξιολόγηση θα έχει αίσιο πέρας και ότι θα μπορέσετε να συμμετέχετε όσο το δυνατόν συντομότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κόλλιο. Κυρία Σκοφιέ, ευχαριστώ πρόεδρε. Να απαντήσω κατά κύριο λόγο σε μία παρατήρηση, αλλά να πω εφ' ότι πραγματικά μου φαίνεται μεταξύ των υπολείπων προσκεκλημένων ότι και η ΜΕΝ και η ΔΕ έχουμε πεγραμμίσει επανειλημμένω ότι οι πολίτε είναι στην καρδιά τη όλη μέρημνα τους Σέγγεν και τη Ευρώπη. Αυτό είναι και η θεμελιώδη αξία ε, και αρχή μας να διασφαλίσουμε, να εξασφαλίσουμε και να ε, προστατεύσουμε τον πολίτη εντός του χώρου αυτού. Αυτό είναι το βασικό μας μήνυμα. Τώρα θα αποπειραθώ να σας παρουσιάσω τη θέση του κράτους της Γαλλίας σε σχέση με τα πρόσφατα γεγονότα που αναφέρατε, τα οποία πραγματικά νομίζω δυσαρέστησαν, στενοχώρησαν πολλές από τις φίλες χώρες. Ίσως να μην έγιναν και κατανοητά και να μην ε, παρουσιάστηκαν και με το σωστό τρόπο και τις σωστές εκφράσεις. Να πω ότι σήμερα στη Γαλλία ε, ανακαλύψαμε ότι Υπάρχουν 11.000 πολίτες, ένας τέταρτος κόσμος, οι οποίοι ζουν σε συνθήκες ε, ένδυας και εξαθλίωσης πολύ δυσάρεστες. Μιλάμε για κοινότητες οι οποίες στις χώρες τους είναι επίσης θύματα διακριτικής μεταχείρισης. Εκεί λοιπόν κάναμε μια ιδιαίτερη προσπάθεια για να τους ενσωματώσουμε καλύτερα. Όμως ε, η όλη κατάσταση έχει και ευρωπαϊκές διαστάσεις, είναι προφανές. Να υπογραμμίσω ότι η κυβέρνησή μας δεν εφίστη προσπαθειών εδώ και πολλούς μήνες, για να μην πω και για περισσότερο διάστημα, εφόσον επανειλημμένως απεσταλμένοι μας πήγαν στο Βουκουρέστι και συνήντησαν τον ε, Ρουμάνο Υπουργό ε, υπεύθυνο για την ενσωμάτωση των Ρωμά στην Ρουμανία. Θεωρήσαμε και είδαμε έτσι ότι η Ρουμανία δεσμεύεται να ε, συνεργαστεί με την αστυνομία του Δήμου του Παρισιού ε, όπου απέστειλε τέσσερις ε, υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται για την εξάρθρωση συστήματος, δικτύου μάλλον εμπορίας ανθρώπων. Υπάρχει συνεργασία λοιπόν με πρώτη μας κυρία, κυρίαρχη μέρημνα να εξασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια σε αυτούς τους ευάλωτους πληθυσμούς. Η Γαλλία λοιπόν έθιξε τα σημεία αυτά επανειλημμένος και μάλιστα προσφάτως. Πιστεύω λοιπόν και η κυβέρνηση το είπε αυτό με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα ότι θέλει να ε, υλοποιεί πλήρως το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ίσως υπήρξαν κάποιες αδεξιότητες στην έκφραση και θα με συγχωρήσετε να μην ε, ξεπεράσω κάποια όρια. Κατάλαβα όμως το μήνυμά σας, το καταγράφω και να είστε βέβαιοι ότι θα το παραπέμψω. Παρόλα αυτά, σήμερα κάθε κράτος μέλος έχει το προνόμιο να προβλέπει τα δικά του μέτρα για το σεβασμό του δικαίου και να, θα πρέπει τα κράτη προέλευση να αναλαμβάνουν τι δικέ του τι ευθύνε ενώπιον των δικών του πολιτών. Η ελευθερία κυκλοφορία των πολιτών που ε, προστατεύεται στο άρθρο 3 του, της συνθήκης δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει κανεί του πολίτε του που ζουν σε συνθήκε επισφαλή σε ένα γειτονικό κράτο, αλλά πραγματικά προσπαθεί να του εξασφαλίσει την ε, αληθινή αξιοπρέπεια. Οι δράσει λοιπόν που ανέλαβε το γαλλικό κράτο νομίζω ότι διεξήχθησαν σε καλό συντονισμό, σε συνθήκε καλή συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα κράτη. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε αρκετά γενναιόδοροι στο μέλλον για να ξεχάσουμε τα δυσάρεστα. Άλλωστε, στα επόμενα στάδια, ε, προφανώς η γαλλική κυβέρνηση θα δώσει ιδιαίτερη σημασία στο να βοηθήσει ε, έμπρακτα όσους χρειάζονται βοήθεια και γι' αυτό ανακοινώθηκε και ένα κοινό πρόγραμμα με χρηματοδότηση ακριβώς για αυτές τις δράσεις όπου η γαλλική κυβέρνηση θα ελέγχει, θα επαληθεύει το κατά πόσον κάθε δαπάνη, το κάθε κονδύλι θα φτάνει στα χέρια αυτών για τους οποίους προορίζεται οι ενδιαφερόμενοι πληθυσμοί πραγματικά να έχουν τις συνθήκες αξιοπρέπειας που τους αξίζουν. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε όλους. Τα καταφέραμε και μάλιστα στην ώρα μας. Ολοκληρώσαμε τους δύο γύρους ομιλητών που προγραμματίζονταν για το πρωί. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο τελικό μέρος της δημερίδας μας. Καταληκτικές παρατηρήσεις. Γι' αυτό θα καλέσω στο βήμα την κυρία Όλγα Δίρεν, γερουσιαστή από το Βέλγιο, την Βελγική Γερουσία, ώστε να ξεκινήσει το τελευταίο τμήμα της συζήτησης. Σας ευχαριστώ όλους.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 και πάλι, σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. To σας παρακαλώ καθίστε για να προλάβουμε το τελευταίο κομμάτι του σεμιναριού μας. Είναι η τελευταία συζήτηση του σεμιναρίου αυτού. Οι βουλευτές που το επιθυμούν μπορούν να πάρουν το λόγο μετά από τους δύο γύρους συμπερασμάτων που θα ακούσουμε. Πρώτα θα συνοψίσω εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να ολοκληρώσω ώστε να προλάβουμε και να μπορείτε να αποχωρησετε γερος εγκαίρως, διότι ξέρω ότι έρχεστε από πολλά διαφορετικά κράτη-μέλη. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου που είχα τη χαρά και την τιμή να προεδρεύσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Διακοινοβουλευτική Επιτροπή κατά την κοινή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωβουλευτών. Το τελευταίο αυτό κομμάτι της συνεδρίασης δεν έχει στόχο να ξανανοίξει τη συζήτηση ή να προσθέσει νέα στοιχεία, διότι νομίζω ότι Ακούσαμε πολλά πράγματα, σε... ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και επικοδομητική η συζήτηση. Θα ήθελα να συνοψίσω τη συζήτηση και να μοιραστώ μαζί σας την δική μου κατανόηση αυτού του νέου ε, πλαισίου στο οποίο ενεργούμε αυτή τη στιγμή. Γράφουμε νέο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής ιστορίας. Πιστεύω ότι ε, το βασικό βήμα είναι η θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, ο, ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης που δημιουργήθηκε πρώτη φορά στο Αμστερντάμ το 1997 έχει γίνει ένας ανεξάρτητος πλήρης ευρωπαϊκός στόχος. και έχει να κάνει με τη ε, διάδραση ανάμεσα στο εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια και, στα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διατηρήσουμε την ε, ελευθερία, την ασφάλεια και δικαιοσύνη ε, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι σημαντικό στοιχείο ε, αυτού του πλαισίου. Έχουμε τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που, απο, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συνθήκης της Λισαβόνας το οποίο ποτέ δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, ποτέ δεν πρέπει να το παραβλέψουμε. Η συνθήκη της Λισαβόνας δεν αποτελεί μόνο ενοποιημένη εκδοχή των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνει και τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων που τώρα έχει γίνει νομικά δεσμευτικός και θέτει τους πολίτες στην καρδιά του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η δημοκρατική λογοδοσία στο μέλλον θα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για να όχι μόνο νομιμοποιεί περισσότερο και να κάνει πιο αποτελεσματικές τις ε, πράξεις μας. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δουλέψουμε σωστά, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που ενισχύουν τη σχέση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε στενά. Ο διάλογος αυτός ήταν απαραίτητος για τον ορισμό της ε, στρατηγικής ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φορείς που συνδέονται με το έργο αυτό, ιδιαίτερα ο ΚΟΖΗ, θα πρέπει να συμπληρώνουν τις εθνικές στρατηγικές ασφαλείας. Είναι σημαντικό αυτό κατά τη δημιουργία νομοθεσίας στην Ευρώπη. Γι' αυτό χαιρετίζουμε κάθε συνεισφορά που έγινε στην διήμερη αυτή η συζήτηση. Πολλά στοιχεία έχουν σημειωθεί και θα πρέπει να συζητηθούν, όπως άλλωστε έγινε κατά τη διάρκεια αυτού του διημέρου. Η συζήτηση αυτή μας έδειξε επίσης ότι μπαίνουμε σε νέα φάση της επιχειρησιακής συνεργασίας. Όσον αφορά τον ε, τις ε, υπηρεσίες που συμμετέχουν στη δημιουργία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Είναι απαραίτητα εργαλεία, ωστόσο οι δράσει των φορέων αυτών θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια μιας στρατηγικής ε, όπου θα αποφεύγεται κάθε επικάλυψη εργασιών. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να υποφελείται. Είναι λοιπόν σημαντικό για την επιχειρησιακή συνεργασία να πραγματοποιείται κάτω από κοινοβουλευτική εποπτεία σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τα δύο αυτά επίπεδα θα πρέπει να λειτουργούν σωστά. Η Κομισιόν θα πρέπει να επιταχύνει την ε, διαδικασία προσαρμογής ε, των υπηρεσιών αυτών στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Οι νομοθε... σχετικές νομοθετικές προτάσεις θα πρέπει λοιπόν να είναι έτοιμες πριν το τέλος του 2011, δύο χρόνια δηλαδή μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Ξέρουμε ότι πραγματοποιούνται οι διαπραγματεύσεις, δεν θα είναι εύκολη δουλειά, αλλά η Επιτροπή σκοπεύει να ολοκληρώσει την διαπραγμάτευση του κειμένου αυτού τον Μάιο του 2013. Ξέρετε ότι δίδεται πενταετής προθεσμία για την προσαρμογή των θεμάτων του προηγούμενου, του πρώην τρίτου πυλώνα. Ε, δεν χρειάζεται όμως να ε, χρησιμοποιήσουμε το σύνολο της προθεσμίας αυτής. Ταυτόχρονα καλούμε τα κράτη-μέλη να βρουν πρακτικές λύσεις ε, και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρχει λογοδοσία και για να μπορούμε να ασκούμε τα καθήκοντά μας και στο Ευρωπαϊκό και στα Εθνικά Κοινοβούλια σε συνεργασία με τους πολίτες. Προτείνω λοιπόν όλοι όσοι συμμετείχαν στη διάσκεψη αυτή να κάνουν ό,τι μπορούν για να παραμένουν σε επαφή με τους ε, βουλευτές της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών σε τακτική βάση. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να γίνει μια επόμενη συνάντηση ε, στην επόμενη Ευρωπαϊκή Προεδρία και υπό την ίδια μορφή να εξετάσουμε τι έχει βελτιωθεί και τι πρέπει περαιτέρω να βελτιωθεί. Η τελική μου παρατήρηση λοιπόν είναι ότι πρέπει να προσθέσουμε πολιτική αξία σε όλες τις αξιολογήσεις των φορέων που σχετίζονται με τον χώρο ελευθερίας δικαιοσύνης και ασφάλειας. Η Europol, η Eurojust, η Frontex και οι φορείς ε, του Schengen. Είμαστε κοινοβούλιο εδώ, είμαστε όλοι βουλευτές. Το θέμα που τίθεται είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εκπροσωπούμε τους πολίτες μας. Αυτό είναι σημαντικό βήμα που έχει γίνει με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Και όπως υπόθηκε, το θέμα εδώ δεν αφορά μόνο την εσωτερική αγορά, το ενιαίο νόμισμα. Η επιτυχία της ευρωπαϊκής ιδέας θα εξαρτηθεί εν μέρη από την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Νομίσματος και της ε, εσωτερικής αγοράς, αλλά και από την ε, έννοια του Ευρωπαίου πολίτη και τα δικαιώματά του. Επανειλημμένα, έχει τονιστεί ότι υπάρχει πολύ σύγχυση με το εξή θέμα. Όλοι οι φορεί που σχετίζονται με τον χώρο ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις αρμοδιότητες των κρατών μελών στον τομέα αυτών, θα πρέπει να έχουν συντονιστικό ε, ρόλο. Ε, στόχος δεν είναι να εξαλείψουν τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, αλλά να συνδυάσουν τις ε, εργασίες των κρατών μελών φαίνεται δύσκολο, έχει σημειωθεί όμως σημαντική πρόοδος σε ε, περιορισμένο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά ξεκινήσαν πριν μόλις 25 χρόνια. Το πρώτο βήμα έγινε με τη σύμβαση Schengen που υπέγραψαν αρχικά πέντε κράτη-μέλη. Τώρα αυτή καλύπτει σχεδόν το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ξεπερνάει και τα όρια της ε, και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στο χώρο Σέγγεν. Έχει λοιπόν σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Βέβαια υπάρχει αντίσταση. Αυτό πάντα ήταν πρόβλημα. Εκφράστηκε και σαφώς ε, κατά τη διάρκεια αυτής της διάσκεψης υπάρχει αντίσταση σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό είναι σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αναφέρθηκαν κάποια παραδείγματα, να σας θυμίσω την περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ισαγγελέα. Έγινε υπό την Ισπανική Προεδρία σεμινάριο με θέμα αυτόν τον σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό ο οποίος ε, προβλεπόταν ε, να, να δημιουργηθεί μετά τη θέση ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Διότι ανήκει στην όλη λογική το θέμα αυτό του να λύνουμε προβλήματα από κοινού σε περίπτωση που η λύση μπορεί να προέλθει αποκλειστικά από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν αναφέρεται ότι απαιτείται ε, κοινό ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο. Χρειάζεται όμως σύγκληση. Χρειάζεται η εναρμόνιση των νομικών ενιών, των εμπειριών και των φορέων για να ορίσουμε κάποια κοινά μοτίβα για να μπορέσουμε να ορίσουμε ποιες πράξεις ε, θα πρέπει να διώκονται. Όταν μιλάμε για διασυνοριακό έγκλημα και διασυνοριακές απειλές που ξεπερνάνε τις δυνατότητες των μεμονωμένων κρατών μελών. Η τελική μου παρατήρηση λοιπόν είναι ότι θέλω να τονίσω τη σημασία της στάση μας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι είναι πολύ τομέας δράσης, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Η συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει διευκολύνει τα πράγματα των αντίων. Οι θεσμικές ρυθμίσεις που απαιτούνται ε, με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας είναι πολύ πιο ε, απαιτητικές από πριν. Θα πρέπει να συνεργαστούμε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε τις κοινέ αυτές προσπάθειες να τις κάνουμε ουσιαστικές ώστε να έχουν πρακτικό αποτέλεσμα ως προς τα βήματα που κάνουμε για να ε, εξυπηρετήσουμε τους πολίτες μας. Οι δυσκολίες δεν είναι μόνο τεχνικές, είναι και πολιτικές. Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε ο κόσμος να γνωρίζει και να γνωρίζει καλύτερα τι συμβαίνει εδώ. Χθες και σήμερα είδαμε ότι υπήρξε σύγχυση, υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις. Μερικές φορές θα πρέπει να ξεκαθαρίζουμε μεταξύ μας τι είναι αλήθεια και τι όχι σχετικά με τη συνθήκη της Λισαβόνας, τους θεσμούς ε, για τους οποίους μιλάμε. Τι είναι και τι δεν είναι αλήθεια για τη Frontex, τι ισχύει και τι όχι για το Σέγγεν. Για να ξεκαθαρίσουμε τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα αυτά και να μεταφέρουμε τι γνώσει αυτέ στου πολίτε μα, πολίτες μας, διότι δεν έχουν ιδέα τι γίνεται εδώ μέσα. Θα πρέπει λοιπόν να μεταφέρουμε τι πληροφορίε αυτέ στου πολίτε μα. θα πρέπει να καταβάλουμε κοινέ προσπάθειε για να του δείξουμε ότι μα ενδιαφέρουν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι οι πολίτε τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα και δουλειά μα είναι αυτόν τον πολύπλοκο αστερισμό θεσμικών και κοινοβουλευτικών σχήματων να τον χρησιμοποιήσουμε για να τους εξυπηρετήσουμε καλύτερα. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Όλγα Ζρίχεν που είναι γερουσιαστής στην Βελγική Γερουσία. Αμέσως μετά θα δώσουμε το λόγο για την τελική συζήτηση. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και επιτρέψτε μου ως πρώην Ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ παρόλο που τώρα εργάζομαι στο Ομοσπονδιακό κράτος και σε άλλο επίπεδο εξουσιών στο Βέλγιο επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι τα λόγια σας τα θεωρώ πολύ κέρια εδώ πραγματικά υπάρχει εντύπωση έλλειψης διαφάνειας και μη προβολής όλων των ευρωπαϊκών κανόνων, ιδίω ό,τι αφορά το κομμάτι της ασφάλειας και των δικαιωμάτων των πολιτών. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γνωρίζετε καλά ότι έχουμε αρκετές δυσκολίες στο ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να εντάξουμε στις ευρύτερες προοπτικές μας την εξέλιξη και μετατροπή της επικράτειας και του συνόλου των κανόνων μας και μόνον σε οικονομικό επίπεδο. Αλλά σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την προστασία των ατομικών ελευθεριών είναι προφανές ότι η βούληση, η επιθυμία για διαφάνεια και λογοδοσία δεν θεωρούνται κεκτημένες από τους πολίτες. Μπορούμε βεβαίω να εκφράσουμε ικανοποίηση για το γεγονός ότι επιτέλους καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη να συνδυάσουμε στις προσπάθειές μας ε, το Ευρωκοινοβούλιο και τη δράση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Το θέμα του δημοκρατικού ελέγχου ε, έχει να κάνει και με την αύξηση των δυνατοτήτων, των λειτουργικών δυνατοτήτων ή της Europol και της Eurojust διότι τη στιγμή της δημιουργίας τους ε, και μεταξύ του τι έχουν πετύχει σήμερα βλέπουμε μεγάλη πρόοδο στη δράση των δύο αυτών οργανισμών. Το είπα λοιπόν, ο δημοκρατικός έλεγχος είναι θεμελιώδης και εδώ η Europol πρέπει να παραμείνει και υπεύθυνη και διαφανής ενώπιον των ε, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω του, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του, της Europol θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία προς το Ευρωκοινοβούλιο. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι κάποιες φορές υπάρχει αίσθηση ότι κυριαρχούν οι επιθυμίες των κυβερνήσεων σε σχέση με των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ιδίω ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ε, Europol δεν είναι... Οι κανόνες για τη Europol δεν είναι απόλυτα σαφείς ως αφορά την απονομή των αρμοδοτήτων, τους διορισμούς. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη ελέγχου. Το είχαμε ήδη πει από το 2002 έπρεπε να αναζητήσουμε τα νομικά μέσα, τα θεσμικά εργαλεία, προκειμένου να ασκήσουμε πραγματικό έλεγχο, δημοκρατικό. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι προτάσεις ε, όπως έχουν καταρτιστεί στη συνθήκη της Λισαβόνας δεν ε, αφήνουν περιθώριο για έλεγχο από τα εθνικά κοινοβούλια στη δράση της Europol, παρόλο που υπήρχε αυτή η επιθυμία διότι οι κανόνες που διέπουν την δράση, τη διάρθρωση, τον πεδίο αρμοδιότητας και τις παρεμβάσεις της Europol ορίζουν μεταξύ των δυνατοτήτων ελέγχου της Europol το σε ποιο βαθμό συμμετέχει το Ευρωκοινοβούλιο και ποιο τα εθνικά κοινοβούλια. Όμω το πώ θα διοργανωθούν μεταξύ του τα Ευρωκοινοβούλια με τα εθνικά κοινοβούλια είναι άλλο θέμα. Είπαμε ότι είναι θεμελιώδου σημασία όλα αυτά να γίνουν πιο εύστοχα, πιο αποτελεσματικά, χωρί να ξεχνάμε την έννοια τη πολιτική, να μην περάσουμε σε μια προσέγγιση τεχνοκρατική, αυτοματοποιημένη. Υπάρχει προστιθέμενη αξία η οποία είναι πολιτική εφής και αφορά τα δικαιώματα τα ατομικά αλλά και τη δυνατότητα που διαθέτουμε να προβλέψουμε πρόσβαση για τους πολίτες στις γενικές πληροφορίες και κυρίως στις καλύτερες πληροφορίες. Θέλουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τα Εθνικά Κοινοβούλια που να εμπιστεύονται με τη σειρά τους το Ευρωκοινοβούλιο. Ναι λοιπόν, πρέπει να υπάρχει και δημοσιονομικός έλεγχος. Ο δημοσιονομικός όμως αυτός έλεγχος βρίσκεται στην καρδιά του κοινοβουλευτικού ελέγχου για ορισμένες πτυχές. Σίγουρα όμως ε, απομένει να δούμε σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων και αυτό είναι μια δουλειά που θα πρέπει να γίνει στην ε, περίπτωση του κάθε κοινοβουλίου ξεχωριστά εκτός μικροφώνου. Ε, το ερώτημα λοιπόν είναι το ερώτημα είναι αν πρέπει να δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή με συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Πόσο συχνά θα συνέρχεται αυτή η επιτροπή, ποιε θα είναι οι αρμοδιότητέ τη θα πρέπει σε κάθε συνάντηση να υπάρχει μια εθνική αντιπροσωπεία, μάλλον εκπροσώπηση των εθνικών αντιπροσωπείων στη Europol. Αυτά είναι θέματα που ακόμη πρέπει να συζητηθούν, διότι είναι κρίμα να γίνονται συναντήσει όπω η σημερινή, να φεύγουμε με κάποιε διαπιστώσει και ωραίε ιδέε. και όπω είπε ο συνάδελφο, να ξαναρχόμαστε μετά λέγοντας ότι δεν μπορέσαμε να επιτελέσουμε το μεταξύ πρόοδο. Σε ό,τι αφορά τη Eurojust, Πράγματι το άρθρο 95, 85 συγγνώμη, της βασικής συνθήκης προβλέπει τα κοινοβούλια να συμμετέχουν στην αξιολόγηση δραστηριοτήτων της Eurojust. Βεβαίω το άρθρο 85.1 της Συνθήκης της Λισαβόνας απαιτεί διαφάνεια, αυξημένη διαφάνεια στο ένομο, στην ένομη άσκηση του ποινικού, των ποινικών δικαιωμάτων. Αυτά ορίζονται για το Κοινοβούλιο στα άρθρα 68 και 69, ενώ στο άρθρο 70 προβλέπεται τα εθνικά κοινοβούλια να λαμβάνουν γνώση της αξιολόγησης της Eurojust. Μπορούμε να πούμε ότι τρόπον την έχουμε τα εργαλεία και τα μέσα για να διενεργήσουμε τον έλεγχο αυτών και την σχετική αξιολόγηση. Το επόμενο λοιπόν ερώτημα είναι ποιος από εμά τα Εθνικά Κοινοβούλια θα ζητήσει να δει τους ελέγχους αυτούς, τις αξιολογήσεις, τις εκθέσεις και όταν θα υποβάλλονται στα Εθνικά Κοινοβούλια ποιος εξετάζει το περιεχόμενο. Έχουμε κοινούς ε, τρόπους, διαγράμματα αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Διότι αφού γίνει αξιολόγηση από δική μας πλευράς πρέπει μετά να έχουμε και διάλογο μεταξύ μας για το τι ε, περιμέναμε από τον έλεγχο αυτό. Υπάρχει και η απόφαση του Συμβουλίου που ιδρύει τη Eurojust, η οποία όμω απλώ προβλέπει ενημέρωση του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων για τι δράσει τη Eurojust. Επιτρέψτε μου λοιπόν να επαναλάβω την έκκλησή μου. Να σας πω ότι πρέπει να σκεφτούμε τα εξή θέματα. Δεν θα πρέπει οι διατάξεις του άρθρου 32 της απόφασης του Συμβουλίου του 2002 να παραταθεί, να περιλάβει τα Εθνικά Κοινοβούλια και να επιτρέψει πραγματική αξιολόγηση χειροπιαστή των δράσεων της Eurojust. Δεν θα πρέπει να σχεδιάσουμε ενίσχυση των δυνατοτήτων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Δεν πρέπει να σκεφτούμε για τη Eurojust πως χρειάζεται μια κοινή δομή υπό τη μορφή μιας κοινή επιτροπής λόγου χάρη με όλα τα συμπαρομαρτούντα. Βεβαίως θα επέμενα στο εξής κοινοβουλευτικός έλεγχος σημαίνει έλεγχος από εκλεγμένους ε, αντιπροσώπους του λαού. Οπότε οφείλουμε να διασφαλίσουμε την επιθυμία των πολιτών μας. Εάν, δημιουργηθούν, ε, εάν δημιουργήθηκαν αυτοί οι δύο οργανισμοί, ο σκοπός δεν ήταν να ενισχυθεί απλώς ο έλεγχος των πολιτών, αλλά να διασφαλιστεί για τους πολίτες ότι θα παρακολουθούμε τα της ασφάλειας, τα της προστασίας των δικαιωμάτων τους και ό,τι αφορά την εξασφάλιση των δημοκρατικών ελευθεριών. Σε αυτό που σήμερα ζούμε, ένα τεράστιο κράτος που αποτελείται με τη σειρά από 27 κράτη. Ο δημοκρατικός λοιπόν έλεγχος θα επιμείνω σε αυτό, πρέπει να παραμείνει υπεύθυνο και ιδιαίτερα διαφανής, ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη για το σύνολο των κανόνων μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σιχέν. Και τώρα κάποια λεπτά για να ξεκινήσει μια τελική στη φάση της συζήτηση. Πρώτα, η κυρία Ντετζιρόλαμο από την Κάμερα Διντιπουτάτη της Ιταλίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα ζητήματα που θίξαμε σε αυτή τη συζήτηση σίγουρα θα έχουν πολύ σημαντικές συνέπειες και σε επίπεδο ευρωπαϊκό και στα κάτι μέλη η ελευθερία, η προστασία των πολιτών, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η καταπολέμηση της λαθομετανάστευσης, της τρομοκρατίας, η ενσωμάτωση μειονοτήτων, όλα αυτά είναι θέματα αλληλένδετα. Τα κάτι μέλη ενδεχομένω δεν έχουν μέσα το καθένα μόνο του να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν κοινέ πολιτικέ. Βεβαίω, η Ευρωπαϊκή Ένωση να τρέχει σε οργανισμού όλο και πιο συστηματικά. Αυτό μα φαίνεται καλή ε, ε, πολιτική. Όμω πρέπει να έχουν και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα οι οργανισμοί αυτοί. Δεν αρκεί ένα σύνολο κανόνων και επιθυμία συνεργασία από την πλευρά των εθνικών αρχών. Θεωρώ λοιπόν ότι μετά όπω είπαμε χθε ε, για την Frontex θα πρέπει να εμπνευστούμε από όλα αυτά και για την Eurojust και την Europol. Βεβαίω χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία, περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερη, καλύτερο σχεδιασμό πολιτική για την, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι όνειδος ε, να εκμεταλλευόμαστε τους λαθρομετανάστες, τους ανθρώπους αυτούς που φτάνουν στην ειδική μας επικράτεια έχοντας ζήσει σε συνθήκες εξαθλίωσης. Υπάρχουν όμως χώρες που είναι πιο εκτεθειμένες γεωγραφικά, όπως η Ιταλία, θα πρέπει εδώ σαφώς να υπάρξει πολιτική αλληλεγγύη, λοιπόν από τους ε, ομιλητέ χθε, είτε τα ευρωβουλευτέ είτε Ιταλοί βουλευτέ, ακούσαμε ότι πρέπει πραγματικά το θέμα τη προστασία των δικαιωμάτων να μα απασχολήσει. Επειδή μιλάμε τώρα για θεμελιδιώδη δικαιώματα, η μεταφορά αρμοδιοτήτων από εθνικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να διασφαλιστεί με τα απαραίτητα όργανα και μέσα για τον καθένα από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και θα πρέπει συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα να υπάρχει και λογοδοσία για το τι έχουν πράξει. Νομίζω ότι εδώ η συμμετοχή όλων των ευρωβουλευτών στην, στον πολιτικό σχεδιασμό των οργανισμών αυτών καθώς και η αξιοποίηση όλων των πολιτικών απόψεων που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούν να διασφαλίσουν καλύτερη πολιτική αναχέτηση αλλά και διαχείριση των ζητημάτων που θίξαμε σήμερα και χθε, αλλά και με το πρόγραμμα τη Στοκόλμη, τελευταία συνεδρίαση Προέδρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οδήγησε σε ανάληψη πρωτοβουλειών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα έγγραφο διαβουλεύσεων και προτού γίνουν νομοθετικέ πρωτοβουλίε ε, αναλυθούν μάλλον πολιτικές, ε, νομικές πρωτοβουλίε για τη Eurojust και τη Europol. Ένα τέτοιο έγγραφο συμβουλευτικό θα είναι μια σαφής συμβολή ώστε να αναζητήσουμε μεθόδους εργασία, χειροπιαστούς και πρακτικούς και να αποφύγουμε κατευθύνσεις επικρίσιμες για το πόσο μπορεί να υποφελείται ένα κράτος περισσότερο από ένα άλλο στο χώρο δικαιοσύνης, ασφαλεια και ελευθερίας. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Καρίδης της Βουλής των Ελλήνων παρακαλώ. Κάναμε αυτό το διήμερο, αποτέλεσε μια καλή εμπειρία για όλους μας. Συμφωνώ και εγώ ότι ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση στα σημαντικά θέματα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης είναι ανάγκη να προχωρήσει πιο γρήγορα. Σε πολλές περιπτώσεις καθυστερεί και εμείς και στα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει ε, αυτό να το οθήσουμε όσο μπορούμε. Είναι γεγονός ότι επίσης αυτό το διήμερο δημιουργήθηκαν και κάποιοι μύθοι και αναπτύχθηκαν και κάποια ψεύτικα διλήμματα. Πιστεύουμε και νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι τελικό συμπέρασμα ότι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών θεσμών και μηχανισμών για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών από την παράνομη μετανάστευση, το άσυλο, τη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στην εμπορία των ανθρώπων είναι τόσο αναγκαία όσο από την άλλη μεριά είναι αναγκαία ε, και ο σεβασμός και η περιφρούρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι αξίες πρέπει να πηγαίνουν μαζί και όχι να συγκρούονται. Έχει επίσης σημασία να φύγουμε από την σημερινή αίθουσα κατανοώντας όλοι, μας ότι όλες οι χώρες δεν φέρουν τα ίδια βάρη για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Υπάρχουν χώρες, ε, μίλησε προηγούμενα η συνάδελφος Ιταλίας για τη χώρα της, θέλουμε και εμείς να μιλήσουμε για την Ελλάδα, που σηκώνουν ένα πολύ μεγάλο βάρος και είναι στο μάτι του κυκλώνα σε σχέση με τα προβλήματα της παράνομης μετανάστευσης, του οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών. Εδώ η ευρωπαϊκή και κοινοτική αλληλεγγύη πρέπει να εκφραστεί όχι μόνο στα λόγια, αλλά να πάρει σάρκα και οστά και με γενναία χρηματοδότηση, αλλά και με καθαρές απαντήσεις, πολιτικές απαντήσεις σε προβλήματα που υπάρχουν και που δυστυχώς αυτό το διήμερο δεν απαντήθηκαν και από τους αρμόδιους. Για μας είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία η κατοχήρωση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η καταδίκη των πολιτικών που αναπτύσσει η Τουρκία στο Αιγαίο και στα θαλάσσια αλλά και στον Εύρο στα χερσαία σύνορα και αυτές οι πολιτικές πρέπει να ε, καταδικαστούν από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες εδώ να μην υπάρξει δηλαδή μια επιλεκτική αντιμετώπιση και να υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις γιατί καταπατούν συμφωνίες και κανονισμούς. Ζητούμε την, την αλλαγή του Διβλίνο 2, ζητούμε την ενίσχυση της Frontex και της Europol και θέλω να κλείσω με την εξής παρατήρηση. Όσο οι Ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται απροστάτευτοι, τόσο θα διεγκώνεται και ο ρατσισμός και η ξενοφοβία και τόσο θα διευρύνεται το έλλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών θεσμών. Είναι χρέος σε όλους μας είτε είμαστε βουλευτές από εθνικά κοινοβούλια, είτε, είμαστε ευρω... είτε οι άλλοι συνάδελφοι ευρωβουλευτές, αυτό το χάσμα που δημιουργείται και που φαίνεται σε όλες τις έρευνες που διεξάγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να το κλείσουμε με συγκεκριμένες απαντήσεις, να προσφέρουμε ασφάλεια στους Ευρωπαίους πολίτες και κυρίως στα θέματα της καθημερινότητάς Γιατί και εγώ, κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ μαζί σας ότι δεν, πρέπει να μας αφορά μόνο το ευρωπαϊκό νόμισμα και οι κοινέ πολιτικές π.χ. στα αγροτικά θέματα, αλλά κυρίως πρέπει να ενισχύσουμε τις πολιτικές εκείνες που αφορούν την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Señora de ευχαριστώ κυρία Γκόμες της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ Πολιτικών Ελευθερών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση ήταν χρήσιμη και πρέπει να συνεχίσουμε αυτά τα οποία ε, αρθρώνει ως λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού με τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίσω κάτι, ότι από τη συζήτηση αυτές τις μέρες κατέστη σαφές πλέον ότι Πολλές πρόοδοι ήδη σημειώθηκαν σε τομείς που κανένας δεν θα το είχε σκεφτεί πριν από 20 χρόνια ότι θα ήταν δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Διότι αφορούσαν τις ε, κυρίαρχες έννοιες των κυρίαρχων δικαιωμάτων των κρατών μας. Γι' αυτό σήμερα είναι θεμελιώδες εμείς ως κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι να καταβάλουμε προσπάθεια να απορρίψουμε αυτού του είδους δικαιολογίες για να παρακολουθούν άλλες πρόοδοι που είναι απόλυτα απαραίτητες όμως και αυτές ε, για να υλοποιήσουμε τις ευθύνες μας για να διασφαλίσουμε την ελευθερία και την ασφάλεια στους πολίτες, στους Ευρωπαίους πολίτες και ένα από αυτά, μία από αυτές τις ανάγκες αδιαμφισβήτητα είναι εκείνη ενός εισαγγελέα, Ευρωπαίου εισαγγελέα για θέματα δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζούμε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης. Ζούμε σε μια εποχή όπου το έγκλημα είναι διεθνικού χαρακτήρα. Παίρνει παγκόσμιες συνιστώσεις και εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία και παίρνει και τις πιο διαφορετικές μορφές και πρόσωπα και χωρίς αυτό το μέσο της εισαγγελίας που είναι προφανώς ότι είναι αναγκαίο για να συμπληρωθούν αυτά τα μέσα που υπάρχουν από πλευρά δικαστικών συστημάτων στα κράτη-μέλη χωρίς την εισαγγελία αυτή η ευρωπαϊκού χαρακτήρα δεν θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την δικαιοσύνη που επιθυμούμε να διασφαλίσουμε για τους πολίτες μας. Πριν από λίγο Είχαμε και το θέμα Σέγγεν το οποίο συζητήσαμε και ο Ευρωβουλευτής Κάρλος Κοέλιο είπε ότι συχνά υπάρχει εντύπωση ότι προστατεύουμε τους πολίτες μας από το εξωτερικό, από τους εξωτερικούς κινδύνους που προέρχονται από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έτσι υποβαθμίζουμε τους κινδύνους που υπάρχουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ υπάρχει ανάγκη ακριβώς ε, της ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για αυτούς τους κινδύνους εκ των έσω, εκ των ένδων, για τους οποίους κινδύνους η, εθνικές ε, η εθνική δικαιοσύνη των κρατών μελών δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνη της. Χρειάζεται μια διεθνή συνεργασία. Εδώ πιστεύω ο ρόλος μας ως Ευρωβουλευτών δεν είναι μόνο να ασκήσουμε αντιμετωπίσουμε τον έλεγχο ή το oversight, την εποπτεία, αλλά να αντιμετωπίσουμε και να νικήσουμε, υπερνικήσουμε τις αντιστάσεις και δισταγμούς εκείνων των κυβερνήσεων και πολιτικών δυνάμεων ή ακόμα και εγκληματικών δυνάμεων που πραγματικά δεν επιθυμούν να έχουμε στα χέρια μας ένα τέτοιο αποτελεσματικό μέσο όπως της εισαγγελία σε αυτή την εποχή στην οποία ζούμε. Δηλαδή το μέσο της Ευρωπαϊκής εισαγγελία στη συνεργασία μας. Και έτσι όπως η Ευρωπόλ, η Eurojust, το Frontex και στο πλαίσιο Schengen μπορούμε να αρθρώσουμε ένα λόγο και να συνεργαστούμε μεταξύ εθνικών αρχών και ευρωπαϊκών αρχών έτσι λοιπόν μπορούμε να προσθέσουμε και να διευρύνουμε κάθε μια από αυτές ε, με το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Πιοτρόβιτς από την Πολωνική Γερουσία. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. άκουσα προσεκτικά μια ολόκληρη σειρά ε, από πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις από τους αγορητές στη συζήτηση που είχαμε αυτές τις μέρες. Και χωρίς αμφιβολία, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται σημαντικά θεσμικά όργανα για να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Αυτό είναι εύλογο και κατανοητό. Όμως χρειάζεται από την άλλη πλευρά να είμαστε και προσεκτικοί, διότι η διοίκηση και η γραφειοκρατία όλο και αυξάνονται και τείνουν να αυξάνονται διότι αυτή είναι η τάση τους. Εδώ χρειάζεται να είμαστε πραγματικά, να βρούμε τη χρυσή τομή. Έχω επιφυλάξεις να δημιουργήσουμε το όργανο του ε, εισαγγελέα. Και αυτό γιατί ένα θεσμικό όργανο χωρίς νομικά μέσα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Είναι πιο σημαντικό λοιπόν πιστεύω εγώ προσωπικά να χρησιμοποιήσουμε τα υφιστάμενα θεσμικά όργανα σωστά, αντί να χρησιμοποιήσουμε νέα θεσμικά όργανα τα οποία θα εγκαθιδρύσουμε, θα συστήσουμε. Και γι' αυτό πρέπει να λάβουμε μέτρα για να διευρυνθεί η αποτελεσματικότητα και η συνεργασία μεταξύ εθνικών εισαγγελικών αρχών και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συνεργασία τους. Ξέρω εμπειρικά ότι υπάρχουν ελλείψεις και κενά σε αυτό τον τομέα. Για παράδειγμα, της νομικής συνδρομής την αρρωγή αυτή μεταξύ των εθνικών, των υπηρεσιών των εθνικών εισαγγελέων. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες, να μην δημιουργήσουμε νέα θεσμικά όργανα, να χρησιμοποιήσουμε τα θεσμικά όργανα τα οποία υφίστανται ήδη για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, διότι φοβούμε ότι η υπερβολική γραφειοκρατία θα βλάψει τη συνεργασία μας. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Κύριο Ντίθε Μέρα από την ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε μία-δύο πρώτα λόγια για να αξιολογήσω με πολύ θετικό τρόπο κιόλα ε, τις δύο αυτές ε, συνόψεις ή περιλήψεις που έγιναν από πλευράς ε, της Προεδρίας. Θα ήθελα να υποβάλω μια πρόταση υποβάλλοντας μια πρόταση που θα ήθελα να συζητηθεί και να αναπτυχθεί στο μέλλον για το, την διαδικασία ελέγχου αυτών των υπηρεσιών και οργανισμών. Φυσικά το πιο λειτουργικό θα ήταν οι διαστάσεις το πλαίσιο το οποίο ήδη ε, παρουσιάσαμε όταν συζητήθηκε η απόφαση του Συμβουλίου που έκανε λόγο για μια μεικτή επιτροπή μεταξύ, το είπε και η εκπρόσωπος της Γερουσίας μεταξύ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτή η μεικτή επιτροπή θα μπορούσε να λειτουργήσει πλήρως ή ε, ε εν μέρη. Η συχνότητα λοιπόν κατά την οποία θα συνερχόταν ετήσια θα πρέπει να είναι αναγκαία ώστε να αντιμετωπιστούν ε, και τα έκτακτα συμβάντα επιπλέον. Έδρα Βρυξέλλες. Το περιεχόμενο και το ουσιαστικό τους πλαίσιο θα ήταν ο προϋπολογισμός που θα είχαν το τμήμα του προϋπολογισμού που θα τα αφορούσε, θα αφορούσε και την η εκτέλεση του προϋπολογισμού που θα αφορούσε αυτά τα όργανα. Δεύτερον, αντικείμενο ελέγχου, οι αιτήσεις δραστηριότητες, εξίσου πάλι προς τις δύο κατευθύνσεις. Η πρόταση δραστηριοτήτων και η εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων. Τρίτο πλαίσιο, διορισμοί. Διορισμοί και πάσεις γενικών διευθυντών και προέδρων των υπηρεσιών και οργανισμών. Και τέταρτο και τελευταίο, θα ερχόντουσαν οι παρουσίες για τον έλεγχο ή παρουσίες για πληροφόρηση από πλευράς τους σε εμά για να γίνεται λόγος και για τα έκτακτα γεγονότα ή ξεχωριστά γεγονότα και έτσι, ολοκληρώνω, θα έπρεπε να εξετάσουμε τον έλεγχο για να υπάρχει πληροφόρηση για αυτά τα γεγονότα μετά από έτοιμα, ίδιο έτοιμα των αρμοδίων των υπηρεσιών αυτών. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Gracias. Σας ευχαριστούμε. Κύριε, κυρία Αλφάνο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε επίσης για το γεγονός ότι αναλάβατε την πρωτοβουλία διοργάνωσης αυτού του σεμιναρίου. Γιατί με αυτόν τον τρόπο τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν την δυνατότητα που τους προσφέρεται να κατανοήσουν καλύτερα με τι ασχολούμαστε εμείς. Ε, έτσι μπόρεσαν και κάποιες αμφιβολίες να αντιμετωπιστούν. Κάνατε λόγο για κάποια σύγχυση που καμιά φορά υπάρχει που κατέστησε σαφές όσον αφορά ρόλους και αρμοδιότητες. Αυτό στις δύο αυτές οι ημερίδες, καταδείχτηκε μεταξύ άλλων. Τώρα, θεωρώ ότι καταδείχθηκε αυτό και πάλι μετά από τα λόγια της Ιταλίδας εκπροσώπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει, σε αντίθεση με τα εθνικά κοινοβούλια, δεν χρειάζεται να δίνει λογαριασμού έναντι των διαφορετικών πρωθυπουργών. Εμεί είμαστε υπεύθυνοι έναντι 500 εκατομμυρίων πολιτών και όχι έναντι κάποιου πρωθυπουργού. Υπάρχουν λοιπόν κράτη-μέλη τα οποία έχουν συμφωνι... Ε, φιλικές, ε, ε, τις φιλικές συμφωνίες τις συγχαίων με συμβάσεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέτοια θέματα τα εντάσσουμε εμείς στις δραστηριότητές μας. Εμείς στην Επιτροπή μας έχουμε για παράδειγμα παρακολουθήσαμε τα, την υπόθεση Ιταλίας-Λιβύης εκ του πρόσφατα και παρακολουθούμε και στο Συμβούλιο το τι γίνεται με τη Λιβύη. Πολλέ φορέ διαπιστώσαμε ότι είναι δύσκολο να παίρνουμε πληροφορίε για αυτή τη, μια τέτοια συμφωνία. Αυτή η Κοινοβουλευτική Επιτροπή βρίσκεται σε εγρήγορση και παρακολουθεί αυτά τα πράγματα. Εκφράσαμε την ε, επιφύλαξή μας και την ε, πραγματικά την αποξένωση που μας δημιούργησε μια, αυτή η συμφωνία. Πρέπει να πούμε ότι κάποια πράγματα δεν πάνε σωστά σε σχέση με κράτη-μέλη. Αυτό δεν έχει σχέση με το ότι εμείς θέλουμε να αυτοδυσφημιστούμε, αλλά επειδή πρέπει να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας. Περνάμε στο τελικό ε, τμήμα αυτής της ε, συνεδρίασης. Δεν βλέπω κάποιοι να έχουν ζητήσει τον λόγο, δεν βλέπω να ζητούν να παρέμβουν κάποια μέλη. Ορθό είναι λοιπόν να προχωρήσουμε στα τελικά συμπεράσματα που θα διατυπώσουν ε, από πλευράς ε, του Προεδρείου οι εκπρόσωποι. Πρώτα απ' όλα από πλευράς μου. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι στόχος μου δεν ήταν να απαντήσω ή να άρω κάποιες ε, παρατηρήσεις που έγιναν σε σχέση με τα όσα ακούσαμε. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων σίγουρα αυτή που είχαμε και ήταν κάτι που μας εμπλούτησε αμοιβαία εσάς και εμάς και μας διαφώτισε και μας ε, ε, αποσαφήνισε πολλά πράγματα για τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν. Όλοι σημειώσαμε κάθε παρέμβαση που ακούστηκε και ελπίζω ότι όλο αυτό το υλικό, όλα αυτά τα στοιχεία θα είναι χρήσιμα κατά κάποιο τρόπο και θα ε, βρουν απήχηση στη δουλειά μας όταν θα στραφούμε πάλι σε αυτήν στα εθνικά κοινοβούλια ή εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο μας για να επεξεργαστούμε και να αφομοιώσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες όλα αυτά τα στοιχεία αξιολόγησης και ανάλυσης για να μπορέσουμε να δουλέψουμε καλύτερα σε αυτό τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε αλλά απλά και μόνο για να συνοψίσω και να ανακεφαλαιώσω κάποια πράγματα κάποια από έλεγα τα στοιχεία αυτά θα ήθελα να πω ότι επανειλημμένα τονίστηκαν από πολλά μέλη, από πολλούς βουλευτές, ιδιαίτερα σε αυτό το τμήμα της συζήτησης. Και θα ήθελα να πω τα εξής. Πρώτον, η σημασία του παράγοντα χρόνου. Ο παράγοντας χρόνος είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα Μάλιστα, καταφέραμε σε ένα σύντομο χρονικό, σε μια σύντομη χρονική περίοδο να σημειώσουμε μεγάλη πρόοδο. Κάποια θεσμικά όργανα τα οποία δεν υπήρχαν πριν από κάμποσα χρόνια, όπως η Frontex, τώρα υπάρχουν και λειτουργούν. Είναι καλό αυτό και θα συνεχίσουν να υφίστανται και να λειτουργούν. Και αυτό έχει κάνει τη διαφορά μεγάλη διαφορά. Έχουν δοθεί παραδείγματα φυσικά και αυτό είναι φυσικό και δεν είναι τυχαίο ότι όταν έχετε η ώρα συζήτηση των Frontex, των θεμάτων Frontex, ακούγονται φωνές από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Μάλτα. Πιο συχνά κιόλα από ότι οι φωνέ από τη Σκανδιναβία. Αυτό είναι απόλυτα φυσικό λόγω τη υφή τη φύση των πραγμάτων. Όμω, γεγονό είναι ότι πριν από λίγα χρόνια, πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχε η Frontex. Δημιουργήθηκε το 2004. Ξεκίνησε τα πρώτα τη βήματα το 2005. Έκανε τη διαφορά, τη μεγάλη διαφορά. Και για τα Κανάρια νησιά, για παράδειγμα, για εμά του ίδιου, μπορούμε να το πούμε αυτό. Ήταν αποφασιστικό αυτό ω στοιχείο. Ενώ μπορεί να υπάρχει κάποια δυσφορία, δυσαρέσκεια όσον αφορά επανειλημμένες ροές ε, ε, μεταναστευτικών ρευμάτων, παράνομων μεταναστών με σκαφίδια, με πλοιάρια. Όμως πρόοδος έχει γίνει παρόλα αυτά και ο χρόνος ε, δεν είναι απεριόριστος. Έχουμε ένα πενταετή περίοδο για τη Λισαβόνα, έτσι δεν είναι μια πενταετή περίοδο για να αναβαθμίσουμε, να επικαιροποιήσουμε την εντολή για την Frontex, την Europol και πρέπει να τα πάμε καλύτερα ώστε να αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποχρεωθεί να κάνει αυτή τη δουλειά έγκαιρα και να σημειωθεί σημαντική πρόοδος για να υλοποιηθούν οι σημαντικοί στόχοι που έχουν εμπλαισιωθεί και έχουν τοποθετηθεί στις διατάξεις της Λισαβόνας και στα όσα προβλέπονται από τις συνθήκες της Λισαβόνας. Το δεύτερο, ενώ περνάει ο καιρός, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο με τα μέσα και τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας τώρα. Να τονίσουμε τη σημασία της αλληλεγγύης και να είμαστε αλληλέγγυοι. Η αναλογικότητα είναι σημαντικό στοιχείο. Η αλληλεγγύη που πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτή που δείχνουμε ενώ είναι περιορισμένη όταν πολλές φορές ε, έρχεται η ώρα να βοηθήσουμε κράτη-μέλη που καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζοντας έκτακτες περιστάσεις. Η Ελλάδα ήταν μια τέτοια περίπτωση επανειλημμένα στο παρελθόν. Θα πρέπει να εξαναγκάσουμε λοιπόν την, ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα το Συμβούλιο, να είναι αλληλέγγυο, να εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους όσους έχουν ανάγκη, διότι αυτό είναι μια θεμελιώδη αρχή για τη διασφάλιση της ε, ε, του χώρου ελευθερίας, ε, ασφάλειας, δικαιοσύνης. Και τώρα για την εξωτερική διάσταση αυτό είναι ένας πυλώνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έχει κατοχυρωθεί στη συνθήκη και αυτό προβλέπεται. Ήρθε επιτέλους η χρονική στιγμή να μάθουμε και να αποδείξουμε ότι ισχύει και βρίσκεται σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Τα κράτη-μέλη το κατέστησαν σαφές και δυνατό μέσω των ε, ε κυβερνήσεων, μέσω του Συμβουλίου να λειτουργήσει αυτό. Και θα πρέπει να συμμορφωθούν τα κράτη-μέλη και οι κυβερνήσεις με τις ίδιες τις τις δεσμεύσεις τους και να εμπλακούν ώστε να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι όλοι. Θα έλεγα επιπλέον ότι Προσέξτε, ένα τελευταίο σημείο που αφορά τις σημαντικές συνεισφορές και παρεμβάσεις που έχουν γίνει για να βελτιωθεί η απόδοση και η ε, δυνατότητα των θεσμικών οργάνων και των υπηρεσιών και οργανισμών. Πολλές προτάσεις ε, έχουν διατυπωθεί πρακτικού χαρακτήρα που έχουν νόημα και έχουν ουσία, ουσιώδης. Σήμερα το πρωί ακούστηκαν πώς μπορούν να βελτιωθούν αυτοί οι οργανισμοί και τα όργανα αυτά. Κάτι που πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως είναι ότι εμεί είμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια που εμπλεκόμαστε άμεσα στην διαρκή εποπτεία, στον έλεγχο για να διασφαλιστεί διαφάνεια, λογοδοσία και το πιο σημαντικό νομιμοποίηση, να νομιμοποιούμεθα έναντι των πολιτών μας με τις δράσεις μας αυτές και την προσπάθειά μας. Αυτό είναι μια διαρκή σε εξέλιξη διαδικασία. Βήμα προς βήμα πρέπει να συνεχίσουμε και να τα καταφέρουμε. Πρέπει να μπορέσουμε να εκπαιδευτούμε σωστά για να αποδώσουμε σωστά. Και ένα πολιτικό συμπέρασμα που θα είναι και η κατακλίδα μου πολιτικό συμπέρασμα. Αν δεν τα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, ο κίνδυνος που διαφαίνεται και διαγράφεται είναι ο λαϊκισμός, η ξενοφοβία, ο φόβος, η φοβία, η πολιτική του φόβου των φοβιών έναντι του άγνωστου του άγνωστου που χτυπά την πόρτα μας, των ξένων, των αλλοδαπών, των άλλων, των διαφορετικών, της, της αυτό δεν μπορεί να είναι η απάντηση. Δεν μπορεί να είναι επιλογή σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Και ο παγκοσμιοποιημένο κόσμο δεν είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει αύριο και θα καταργηθεί. Είναι μόνιμο στοιχείο και χαρακτήρα η παγκοσμιοποίηση. Θα είναι και θα μείνει και πρέπει να το ξέρουμε. Μπορούμε να τα, κάνουμε, να καταφέρουμε πολύ καλύτερα. Αν δεν θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παγιδευτεί σε ένα λόγο ξενοφοβίας και λαϊκισμού, πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες και αν δεν θέλουμε τα εθνικά, η εθνική πολιτική να αντιστραφεί και να έχουμε μια ολόκληρη σειρά εξεγέρσεων και ας το πω έτσι διαμαρτυρίας λαϊκιστικού χαρακτήρα και ρατσιστικής ε, τάσης ε, όπως έχει καταδειχθεί κιόλας ότι σημαίνει, συμβαίνει σε κάποιες εκλογές που έλαβαν χώρα σε κάποια κράτη-μέλη πρόσφατα στη Σουηδία για παράδειγμα και αλλού ε, τότε πιστεύω ότι θα πρέπει να δραθούμε της ευκαιρίας να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν εδώ για την προθυμία τους ε, να υπάρξει αυτή η πληροφόρηση και αυτή η ροή ε, ε, αμφωτέρωθεν και δίνω τώρα τον λόγο για τις τελικές τελευταίες παρατηρήσεις στην συνάδελφο από την Βελγική Γερουσία. Παρακαλώ κυρία Ζήχεν, έχετε τον λόγο. Euh, το όντι, όσα υπόθηκαν είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να συνεχιστεί η όλη προσπάθεια. Ελπίζω ότι θα έχουμε τη χαρά να ξανασυναντηθούμε. Επειδή ξεκινήσαμε εδώ σήμερα, όμω δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει αύριο να προσπαθήσουμε αλλού. Παρακαλώ λοιπόν αυτό το ντοσιέ μην το βάλετε στο κάτω μέρο τη στίβα σα. Να γίνει ντοσιέ προτεραιότητα το θέμα. Όλους μας ε, αφορά Είδαμε ότι όλοι ζήτησαν το λόγο, πολλοί ήθελαν να συμμετέχουν και ξέρετε ότι αξιολογούμαστε με γνώμονα και μέτρο το πόση δουλειά κάνουμε και το τι δουλειά κάνουμε για όλα τα κράτη και τους πολίτες μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και πραγματικά συνεχίστε το έργο που ξεκίνησε η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έρθουμε σύντομα πάλι εδώ με προτάσεις. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους. Γεια σας.